Καλημέρα σας. Θα έλεγα συνάδελφοι, αλλά μάλλον είναι στον ενικό συνάδελφε, γιατί είναι έκτακτη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δυστυχώς πολλές πολιτικές ομάδες οργανώνουν τις ημερίδες τους εκτός Βρυξελών. Ελπίζω πάντως, έστω και αργότερα, να έρθουν και άλλοι βουλευτές. Καλή σας μέρα λοιπόν και να καλωσορίσω και την αντιπροσωπεία γηγενών πληθυσμών από την Αφρική. Καλώς ήρθατε. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την αντιπροσωπεία που βρίσκεται συνεδρίε. Έχουμε την κυρία Αϊσά Τομούρου Ιμπραχήμ από τη Δημοκρατία του Τσάτ. Εργάζεται στο, στην Ένωση αυτόχθονων ε, πληθυσμών γυναικών και μάλιστα είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και μάλιστα έχει παρακολουθήσει και κατάρτιση για τη διαχείριση δασών και τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών. Έχουμε διπλέτη την κυρία Σίνα Τμπάλη. Καλημέρα σας. Είναι του ΑΡΕΓ από το Μάλι. <clears throat> Ξέρω ότι έχετε πολύ καλή μουσική. Ακούω πολύ συχνά μουσικά κομμάτια από την πατρίδα σας στο Μάλι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και συναρπαστική. Είναι το αρέκο, που είπα η κυρία Μάλι. Εργάζεται στην Ατσμόρ, που είναι μια ένωση γηγενών κοινοτήτων από τις βόρειες περιοχές του Μάλι. Και έχουμε και τον κύριο Γιώζεφ Ιταουαν Μοκούμο. Είναι πυγμαίος Μαμπούτη. και διαμένει στην ε, Δημοκρατία του Κονγκό. Ασχολείται με θέματα ανάπτυξη πέθρου και προγράμματα ένταξης ε, της κοινότητας των πυγμαίων στο Κίμπου. Θα θέλετε το λόγο για κανένα δύο λεπτά ο καθένας. Α, ξέχασα τον κύριο... Α, ο κύριε Γιώζεφ μου Μήπως θα θέλετε εσείς εκ μέρους ε, της αντιπροσωπείας σας να λάβετε το λόγο. Vous ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε συντάξει μία κοινή δήλωση των τριών εκπροσώπων για να κερδίσουμε και λίγο χρόνο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, μέλη της Υποεπιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Εκπροσωπούμε τις αυτόχθονες κοινότητες, γαλλόφωνες αυτόχθονες κοινότητες από την Αφρική, από το Τσάτ, το Μαλί και την Δημοκρατία του Κονγκό. Σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας δώσατε και την ευκαιρία να λάβουμε το λόγο στη συνεδρίασή σας, επευκαιρία της επίσκεψής μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα πλαίσια του προγράμματος ε, Διαβίβαση τεχνογνωσία από το Κέντρο Τεκμηρίωσης Έρευνας και Πληροφορίας για τους Αυτόχθονες Πληθυσμούς εφαρμόζουμε αυτό το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέλαμε λοιπόν να, ε, να σας παρουσιάσουμε τις ανησυχίες μας σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις κοινότητές μας. Κυρία Πρόεδρε, 250.000 ε, αυτόχθονοι του Τσάτ, που είναι 2,3% του συνολικού πληθυσμού του Τσάτ, είναι νομάδες ε, βοσκοί. Δεν αναγνωρίζονται όμως ω αυτόχθονος ε, λαός και δεν τυχάνουν καμία ιδιαίτερη προσοχή από το κράτος. Παρόλο που βρίσκονται και σε άλλες περιοχέ του κόσμου, οι Πελμορόρο βρίσκονται περισσότερο στην νότια πλευρά του Τσάτ και εκεί αντιμετωπίζουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την κτηνοτροφία, γιατί δεν έχουν αρκετέ κτηνοτροφικέ γέε, ούτε μπορούν να μεταφέρουν ε, για, από τα χυμαριά τα ζώα τους. Και μάλιστα ο νόμος ε, του 1987 έχει περιορίσει τις δυνατότητες διακίνησης αυτού το, αυτής αυτόχθονης κοινότητας ε, και δημιουργεί προβλήματα και με τους γεωργούς. Παρ' όλα αυτά, ο νόμος 4 της 31 Οκτωβρίου του 1959 προβλέπει κάποια προνόμια και αναγνωρίζει το καθεστώς των ομάδων και είχε μάλιστα ρυθμίσει τις κτηνοτροφικές τους δραστηριότητες. Μάλιστα το υγειονομικό και εκπαιδευτικό σύστημα του Τσάντ δεν είναι προσιτό στους αυτόχθονες πληθυσμού, ενώ, στους πληθυσμούς, ενώ η ζωή των γυναικών είναι ιδιαίτερα επισφαλής. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν μια βοήθεια για την κτηνοτροφική τους δραστηριότητα και μια ιδιαίτερη προσοχή από το Τσάντ. Η δημοκρατία του Μαλή είναι από τις χώρες της Δυτικής Αφρικής που έχει και ε, του ΑΡΕΓ, ένας αυτόχθονος λαός που εκμεταλλεύεται εδάφη της Σαχάρας που βρίσκεται στο Μάλι. Βέβαια, κυρίως ε, έχουν εισοδήματα από την κτηνοτροφία και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ξηρασίας ε, και της, του λοιμού. Δυστυχώς οι δραστηριότητε τους δεν τη χάνουν καμίας κοινωνικής προστασίας, καμίας εγγύησης. Χρειάζονται βοήθεια για να καταπολεμήσουν τα προβλήματα της ανομβρίας και να διερευνήσουν εναλλακτικές λύσεις, να καταπολεμήσουν ε, το λοιμό και να προωθήσουν την ε, κοινωνική τους κατάσταση. Θέλουμε κάποια αλλαγή του καθεστώτος ώστε να προστατευτεί η απασχόλησή τους και να θαρρυνθεί η κοινωνική τους ένταξη. Μάλιστα, χρειάζεται μεγαλύτερη αποκέντρωση, ενίσχυση των δικαιωμάτων των ε, ομάδων, και αναγνώριση της ε, κτηνοτροφικής του δραστηριότητα. Αυτό είναι προτεραιότητα για το ΣΤΟΑΡΕΚ. Στο Κογκό έχουμε 600.000 ε, αυτόχθονους, 1% ε, δηλαδή του κογκολέζικου πληθυσμού. Η κοινότητα Μαμπούτη έχει πάνω από 40.000 ε, ανθρώπους στο Κίβου και μάλιστα είναι η ομάδα αυτή μία από τις μεγαλύτερες αυτόχθονες ομάδες. Οι Μαμπούτι έχουν αναγνωριστεί ως αυτόχθονος πληθυσμός και ο, τρόπος, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής τους ε, έχει αναγνωριστεί. Βέβαια, οι εμπόλεμες σειράξεις που ε, έπληξαν τη χώρα έκαναν πιο ευάλωτο τον αυτόχθονο πληθυσμό Μαμπούτη που ούτως ή άλλως ε, χρόνια ολόκληρη ήταν θύματα της αναρχικής ε, εκμετάλλευσης των ε, φυσικών πόρων, των ορυχείων και των δασών που περιορίζουν το ζωτικό τους χώρο και η μη συμμετοχή τους στα όργανα λήψη αποφάσεων καταστρατηγούν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και τα δικαιώματα των αυτόχθων πληθυσμών, όπως το άρθρο 8G τη Σύμβαση για τη Βιοπικιλότητα και τη διακήρυξη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτόχθων πληθυσμών. Κύριε Πρόεδρε, τα αναπτυξιακά προγράμματα και αποκατάσταση της ειρήνης που έχουν ξεκινήσει στο Κονγκό σε συνεργασία με τους εταίρους της, όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ συχνά αυτά τα προγράμματα αγνοούν τα δικαιώματα των Μαμπούτη. Και η συμμετοχή του στο πρόβλημα σταθεροποίησης και ανασυγκρότησης ε, της Δημοκρατίας του Κονγκό, δηλαδή το πρόγραμμα ΣΤΑΡΕΓ, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΙΕ, θα πρέπει να συμπεριλάβει και το λαό Μαμπούτη και να λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα και την ειδική του θέση και στα άλλα προγράμματα και σχέδια που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις περιοχές που κατοικούν. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, θα θέλαμε την παρέμβασή στους ώστε οι περιθωριοποιημένοι αυτόχθονες πληθυσμοί να μπορούν πολύ πιο εύκολα ε, να, να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους και να θεωρηθούν ως προτεραιότητες στις χρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you so much for these words and I... Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Σας διαβεβαιώ ότι η υποεπιτροπή μας ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των αυτοχθών πληθυσμών και γι' αυτό ε, είχαμε και εκπροσώπους ε, στο συνέδριο ε, του ΟΗΕ των εκπροσώπων των αυτοχθών πληθυσμών πέρσι. βλέπω ότι, ότι η επιστημονική διευθυντής των αυτοχθών πληθυσμών ως προς την τεκμηρίωση είναι μαζί μας και θα ήθελε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι βουλευτές. Ήθελα να υπενθυμίσω ότι το πρόγραμμα ενίσχυση των ενδογενών ικανοτήτων των φτωχών πληθυσμών στον ΟΗΕ χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αλλά επίσης υλοποιείται σε εταιρική σχέση με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η υπηρεσία που εκπροσωπώ εδώ και 30 χρόνια συνεργάζεται με τους εκπροσώπους των αυτοχθών πληθυσμών στον ΟΗΕ κατόπιν αιτήματό του συστάθηκε ε, και παρέχει αμερόληπτες ε, υπηρεσίες τεκμηρίως σε τέσσερις γλώσσες, σε κινέζικα και φορές και πορτογαλικά γιατί κάποιοι έρχονται από τη Βραζιλία, υποβάλλουν έτσι τα αιτήματά τους στον ΟΗΕ, έχουν υλικοτεχνική υποστήριξη ε, Στι γενικέ συνελεύσει του ΟΗΕ συνεργαζόμαστε και με την Γραμματεία τη Εμμόνιμης υπηρεσία εκπροσώπηση των Αυτοχών Πληθυσμών στη Νέα Υόρκη. Για να μην μακρηγορώ θα σα έλεγα ε, συνοπτικά ότι κάνουμε ό,τι δεν μπορεί να κάνει ο ΙΕ ούτω ώστε οι αυτόχθονε πληθυσμοί να ε, συμβάλλουν στη διαδικασία ενίσχυση των δικαιωμάτων του Με από πλευρά υλικοτεχνική στηρίξη, συμμετείχαμε και στην δήλωση των δικαιωμάτων αυτοχθόνων πληθυσμών που εγκρίνει ιδρύθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον ΟΗΕ το 2006 και που αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, των γηγενών πληθυσμών. Ε, προφανώς ε, βέβαια όλα αυτά υπάγονται στη Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, του ΟΗΕ. Το 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε το μοναδικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας μας, της ΔΟΣΥΠ. Δεν θέλω να μας κάνω διαφήμιση. Ε, γιατί κανείς δεν το θέλει αυτό, ούτε και οι εκπρόσωποι των γεννών πληθυσμών. Θα έλεγα πάντως ότι έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική στην Γενέβη και δεν θέλουμε να καταχραστούμε τις θέσεις μας, ε, αλλά παρόλα αυτά το 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε την ιδιαιτερότητα των ε, δραστηριοτήτων μας και μας έδωσε ένα συγκεκριμένο στόχο, δηλαδή την χρηματοδότηση κάποιων προγραμμάτων. Τώρα βέβαια μας αρνούνται αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς και μας λένε ότι πρέπει να συνεργαστούμε με μια διακυβερνητική οργάνωση. Αυτό όμω δημιουργεί πρόβλημα ε, ακριβώ ω προ την αμεροληψία των δραστηριοτήτων Μα Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάποιε ανθρωπιστικέ οργανώσει δεν είναι ελεύθερε όπως ε, εμείς, ε, ούτε τόσο, έχουν τόσο μεγάλη κινητικότητα και τόσο μεγάλη ευελιξία όπω η δική μα υπηρεσία. Οπότε ζητούμε εδώ να υποστηρίξετε μια επιχειρηματολογία που έχουμε μοιράσει ήδη στα αγγλικά και στα γαλλικά για να τεκμηριώσουμε, να στοιχειοθετήσουμε αυτό το αίτημά μα, το οποίο υποβάλλει βάλουμε στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, και έγκυται στο εξή. Αν έχετε τη δυνατότητα, θα θέλαμε να εισηγηθείτε μια τροπολογία για την αθεώρηση τη νομική βάση του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τι οργανώσει που υποστηρίζει εξ ορισμού, όπω παραδείγματο χάρη την είπατε, αρμοστία για τα ανθρώπινα δικαιώματα το ΙΕ και να προσθέσετε εκεί την ΤΟΣΥΠ, τη δική μα υπηρεσία. Ε, υπενθυμίζω το 2009 μα υποστηρίξατε ήδη και ανησυχούμε διότι αν χάσουμε τη χρηματοδότηση θα αντιμετωπίσουμε μεγάλες δυσκολίες. Βέβαια από την Ελβετία, από τη Γενέβη λαμβάνουμε κάποια χρηματοδότηση αλλά δεν επαρκεί οπότε δεν μπορέσουμε να στηρίξουμε τους γηγενείς πληθυσμούς, δεν θα μπορούν να εκφράζονται κατά το δέον και μόλις εγκριθεί το ψήφισμα πρέπει και να υλοποιηθεί. Είναι σημαντικό, υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί στο ΝΟΙΟ που μας επιτρέπουν ε, την εποπτεία, την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων. Ε, κάθε φορά που υπάρχουν διαφωνίες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι δυνατή η προσφυγή σε διεθνέ επίπεδο στη δική μα υπηρεσία, στα πλαίσια πάντου του ΟΗΕ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρο. Σημειώνουμε το αίτημά σα και φυσικά εμπλεκόμαστε όλο ιδιαίτερο στη ρύθμιση τη εποπτεία τη χρήση του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και θα εξετάσουμε ε, αυτό το θέμα τώρα. Θα ήθελα να πω καλημέρα συνάδελφοι, γιατί μέχρι στιγμή υπήρχε ένα συνάδελφο. ο κύριο Χάου. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Απλώ, ε, όπω και η Πρόεδρο, θα ήθελα να καλωσορίσω του φίλου ε, και τι ε, συναδέλφου από τον ΤΟΙΣΥΠ. Δεν είμαι ειδικό για το χρηματοδοτικό κανονισμό, αλλά συμφωνώ με αυτό που είπατε. Η κυρία Λοπέζ είναι συνεισηγήτρια για αυτό το θέμα. και Ελπίζω όλοι οι συνάδελφοι εδώ και σκιώδεις εισηγητές να έχουν σημειώσει το αίτημα και ίσως βρούμε κάποιο άλλο τρόπο να παρακάμψουμε το πρόβλημα για να καταγραφεί στα πρακτικά να σα πω ότι στη Γενέβη. Ε, θα θέλαμε να μας δώσετε την ευκαιρία να συζητήσουμε με γηγενείς, με εκπροσώπους των αυτοχθόνων πληθυσμών για να κατανοήσουμε την κατάσταση ε, στα πλαίσια του Ανθρωπιστικού Συμβουλίου και θα, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη μέχρι τούδε συμβολή σας και επίσης ε, να ευχαριστήσω τη συνεισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε για την εξορετική βιομηχανία και τις επιπτώσεις που είχε στους αυτόχθονες πληθυσμούς. Είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα που μας ε, προβληματίζουν. Θα ήθελα να σας συγχαρώ δημοσίως για το έργο σας ε, σε όλους αυτούς τους τομείς μέχρι στιγμή. Σας ευχαριστούμε. Ε, φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη διερμηνία προς τα γαλλικά, λέει η Πρόεδρος. Όχι, διορθώθηκε. ευχαριστούμε κύριε Χάουιτ. Όντω, το Μάρτιο θα στείλουμε κλιμάκιο στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα έχουμε επικαιροποιημένε πληροφορίε για τι δραστηριότητε που σχετίζονται με του γηγενεί πληθυσμού. Θα ήθελα να κάνω κάποιε ανακοινώσει τώρα. Προφανώς το βραβείο των Νόμπελ Ειρήνης πρέπει να το σχολιάσουμε σε διάφορα φόρα στο Κοινοβούλιο. Ο Λίου Ξιαμπό έχει λάβει τα συγχαρητήρια γιατί έλαβε το Νόμπελ Ειρηνή, Είναι ακτιβιστή ε, υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, ο πρόεδρος, ε, ο κύριο Μπουζέκ, είπε ότι όταν υπερασπίζεται κανείς την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα με ειρηνικό τρόπο δεν πρέπει σίγουρα να καταδικάζεται σε εγκλισμό ή σε φυλάκιση και ε, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τα υπερασπιζόμαστε. Η ύπατη εκπρόσωπος, η κυρία Άστον, είπε ότι επιθυμεί ο κύριος Λιουξιαμπό να είναι σε θέση ο ίδιος να μεταβεί και να ε, παραλάβει το βραβείο του. Είναι ένας διπλωματικός τρόπος ε, για να ζητήσει ύπατη εκπρόσωπος την απελευθέρωσή του. Αλλά αυτή είναι η δική μου ερμηνεία. Να σας πω κάτι άλλο που μας ανησυχεί όμως τώρα. Την περασμένη Τετάρτη Έγινε συνέντευξη τύπου, μετά τη συν... ε, ακυρώθηκε συγγνώμη, συνέντευξη τύπου, χωρί κανένα ιδιαίτερο λόγο, μετά τη Σύνοδο Κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα. Υπήρχαν πολλοί λόγοι, ίσω δεν είναι πρόβλημα προγραμματισμού, δεν είχαν αρκετά να πούνε, αλλά πάντω ε, τα γραφεία τύπου ενημερώθηκαν για το ότι κρυβόταν κάτι άλλο πίσω από αυτό. Τέσσερι δημοσιογράφοι από την Κίνα που είχαν τα διαπιστευτήρια ε, για να εισέρχονται στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τελικά παρεμποδίστηκαν και δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν σε αυτή την ε, ανακοινωθήσα συνέντευξη τύπου. Φυσικά υπάρχουν διάφορε εξηγήσει γι' αυτό, αλλά πώ το ερμηνεύω εγώ ότι η λογοκρισία της Κίνας, που είναι γνωστή σε όλους μας, ε, έφτασε και τις Βρυξέλλες και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε να συνεχίσει Εφόσον ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς αποφάσισε για τους ε, τέσσερις ε, δημοσιογράφους, δηλαδή από κινέζικης πλευράς θεωρήθηκαν ως κίνδυνος για την ασφάλεια, αλλά τελικά ήρθαν αυτοί οι τέσσερις δημοσιογράφοι, αλλά παρόλα αυτά ως αντίτιμο αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακυρώσει τη συνέντευξη τύπου. Ο Λίουξ και το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης μας υπενθυμίζουν ότι ε, δεν έχει παρέλθει ο καιρό όπου πρέπει να συζητάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μιλάμε μόνο για στρατηγική ε, συνεργασία, οικονομική συνεργασία, ε, μεταφορά τεχνογνωσίας, αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα που πρέπει να μας απασχολούν. Ο Βέντζι Αμπό, ο πρωθυπουργό ο τι τις περασμένες εβδομάδες πολλάκι αναφέρθηκε στην ανάγκη τη ελευθερία ελευθερίας λόγου, δηλαδή να κατοχυρηθεί το δικαίωμα ε, ε, ε, επικρίσεων από πλευρά του πληθυσμού για τι κυβερνητικέ δραστηριότητε. Γιατί και ο ίδιο έχει πέσει θύμα. Το επίσημο γραφείο τύπου τη Κίνα ε, όταν συνέταξε την έκθεση για την επίσκεψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέλειψε αυτή τη δήλωση που σχετίζεται με την ειδική οικονομική ζώνη που διαπραγματευόμαστε τώρα από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση με την Κίνα. Δεν πρέπει να αφήσουμε σε, με κανέναν τρόπο τη λογοκρισία τη Κίνα να φτάσει στι Βρυξέλλε. Επίσης, κατόπιν αιτήματος ε, του ε, Ανρίκη Αϊνέ, ε, έστειλα επιστολή στον Κινέζο πρέσβη στην Παρατή Ευρωπαϊκή Ενώση για τις ανησυχίες που έχουμε σχετικά με τη μειονότητα Αϊγκουρού στο Σινγκιάνγκ ε, ακτιβιστές, ε, bloggers ε, κατηγορήθηκαν ότι ενεθάρρυναν τη στάση τον Ιούλιο του 2009 Αλή Αντίλ Γελή είναι ο βασι, βασικότερος ακτιβιστής ε, ε, που είναι ο γιος της κυρίας Καγίρα, Καγύρα ε, εκπροσώπου της μειονότητας αυτής, ε, κακοποιήθηκε και υπέστη βασανιστήρια στην Ξινγιάνγκα, στη φυλακή και βάσει διαφορών πηγών έχει επιδεινωθεί τα μάλα η υγεία του. Οπότε τονίζω στην επιστολή μου ότι χρειαζόμαστε πλήρη και μερόληπτη έρευνα για αυτούς τους ισχυρισμούς σχετικά με τα βασανιστήρια του κυρίου Χαλίτιν και ότι θα έπρεπε οι κινέζικες αρχές να προβούν σε αυτήν την έρευνα. Ζήτησε επίσης αναθεώρηση τη υπόθεση της κυρίας Γουν Μίρα Ιμίν ε, που καταδικάστηκε ε, σε φυλάκιση, σόβια φυλάκιση, όταν ε, έγιναν τα επεισόδια το 2009 στην αυτόνομη περιοχή Ξιν Γιάνγκ. Και να σας πω και κάτι άλλο τώρα για τη Ρωσία. Υπάρχουν διάφορες εκθέσει τις τελευταίες εβδομάδες βάσει των οποίων ε, αυξάνονται οι απειλέ ε, ε, προ του εκπροσώπου και υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίω στο Βόρειο Κάφκασο. Θα ήθελα να αναφερθώ στην κυρία Μαγκόμεντοβα, στις 29 Νοεμβρίου η Υποεπιτροπή θα εξετάσει αυτό το θέμα και εν ώψη της διαβούλευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα γίνει στα μέσα Νοεμβρίου με τη Ρωσία θα κάνουμε ένα briefing, μια ενημέρωση πριν τη συνάντηση και ζητούμε λεπτομέρειες σχετικά με την αθεώρηση COHOM για τις διαβουλεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Α, ναι, και ξέχασα ότι οι πολιτικέ ομάδε ε, φαίνεται να έχουν καταλήξει σε συμφωνία βάσει τη οποία την επόμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προετοιμάσει κατεπήγον ψήφισμα για τι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βόρειο Κάφκασο και συγκεκριμένα για την ε, υπόθεση Όλεγ Όρλοφ. Θα θυμάστε ότι ο κύριος Όρλοφ εκπροσωπεί ε, τους νικητές του βραβείου Ζαχάροφ ε, το 2010 γιατί είναι πρόεδρος ε, του Ιδρύματος Memorial και αντιμετωπίζει ποινικέ κατηγορίες από την κυβερνήτη της Τσετσενίας, τον κύριο Κάντιροφ. Είναι απαράδεκτο, είναι ατυχές ο κύριος Όρλεφ να παρεμποδιστεί κατά αυτόν τον τρόπο να μεταβεί την ερχόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο την 21η, διότι αντιμετωπίζει ακριβώς αυτές τις ποινικέ κατηγορίες. Τον προσκαλέσαμε να παρα όταν ο νικητής του βραβείου Ζαχάροβ 2010 θα ανακοινωθεί αφού ληφθεί η σχετική απόφαση. Οπότε ελπίζω συναδελφοί ότι οι πολιτικές ομάδες θα στηρίξουν αυτή την αυτό το επίκαιρο σημαντικό ε, ψήφισμα ε, και νομίζω ότι σήμερα οι ηγέτες των πολιτικών κομμάτων θα αποφασίσουν επ' αυτού. Μία σύντομη αναφορά τώρα ε, για το, την Pride Race στο Βερολίνο. Το... το στο Βελιγράδι. Ε, ε, ε, στις 10 Οκτωβρίου 2.000 άτομα μαζεύτηκαν στο Βερολίνο προς υποστήριξη της Bright Parade. Κάποιοι από εμά συμμετείχαν και ο πρέσβης Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχε και αυτό αποτελεί ενθερμή υποστήριξη ε, Λαμβάνοντα υπόψη και το ψήφιμα, ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των ε, ε, ομοφιλοφίλων και φιλομεταβατικών η κυρία Μαρέα Κορνέλης, επίσης συνάδελφός μας, συμμετείχε στην Παρέιντες στο Βελιγράδι ε, υπήρχε ισχυρότατη αστυνομική παρουσία ενώ οι δρόμοι ήταν άδειοι. Ε, παρόλα αυτά στο Βελιγράδι σε πολλές συνοικίες έγιναν, ε, υπήρξαν ταραχές ανάμεσα σε χούλιγκαν ε, και διαδηλωτές ε, και του, τις αστυνομικές δυνάμεις και τελικά πάνω από 150 τραυματίστηκαν, 250 φυλακίστηκαν, ε, καταστράφηκαν αυτοκίνητα, βιτρίνες ε, ε, καταστημάτων, μεγάλες οικονομικές απώλειες. Ελπίζουμε ότι το Βελιγράδι θα βρει κάποιο τρόπο για να ενισχύσει την ενοχή προς άλλους και ότι αυτά δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Σουδάν τώρα. Θα ήθελα να καλωσορίσουμε θερμά την ε, απόφαση του, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΙΕ σε ό,τι αφορά την εκτολή ανεξάρτητου αμπειρογνώμονα για το Σουδάν που έχει ανανεωθεί. Είναι σημαντικό οι δραστηριότητε του ειδικού επισταλμένου να συνεχιστούν στο Σουδάν, ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη περίοδο που η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν δυστυχώ επιδεινώνεται. Και εν ώψη του δημοψηφίσματος του Ιανουαρίου του 2011 για την αυτοδιάθεση του, του, του νοτιού τμήματος του Σουδάν, η παράταση της εντολής του δικού είναι ακόμη πιο σημαντική. Σε ό,τι αφορά την δημοκρατία του Κονγκό, μετά από την κοινή ακρόση που διοργανώσαμε τον Ιούλιο, το Προεδρείο της Μικτής Κοινοβουλευτικής Συνέλευση αποφάσισε στην επόμενη ε, Ολομέλεια στην Κινσάσα να διοργανώσει μια ειδική συνεδρίαση και χαιρόμαστε για την ε, εξέλιξη αυτή. Ο πρόεδρος Γερουσίας και πολλά μέλη της Κογκολέζικης Βουλής θα συμμετέχουν σε αυτή την ε, επερχόμενη ειδική συνδιάσκεψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο συμπρόεδρος Λουί Μισελ εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε να συμπεριλάβει τα συμπεράσματα της ακρόασής μας στις διμερείς συζητήσεις που θα έχει με τον πρόεδρο Καμπίλα και άλλους οι θύνοντες της κογκολέζικες κυβέρνησης. Μην ξεχνάτε και το ψήφισμα που υιοθετήσαμε για το Δημοκρατία του Κογκό στις 7 Οκτωβρίου στην πρόσφατη Ολομέλεια, όπου επισημαίνουμε τα προβλήματα που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την προσοχή ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την απονομή δικαιοσύνη στη Δημοκρατία του Κογκό. Πλησιάζω προς το τέλος των ανακοινώσεων μου για την Κυριαζία. Μας απασχολεί ιδιαίτερα η κατάσταση του κυρίου Αζημία Ασκάροφ που είναι ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Κυργιζίας και στις 5 Σεπτεμβρίου καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη και δίμευση της περιουσίας του. Ήδη τον Ιούνιο είχα στείλει επιστολή στον πρέσβη της Κυργιζίας επισημένοντας την ανησυχία μου ότι δεν έγιναν σεβαστά τα δικαιώματα δίκαιες δίκης του κυρίου Ασκάροφ που είναι ένας επιφανής ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διευθυντής ε, μιας ε, οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εδρεύει στην κυργεζία. Και μάλιστα συγκέντρωσε, διάφορα στοιχεία για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και διώξεις κατά των Ουσμπέκων Κυργεζίων στα νότια του Κυργεστάν. Και μάλιστα στην περιοχή Νόκεν το Οκτώβριο είχαμε ε, την ε, επανάληψη της δήλωσης ε, να θεωρηθεί η δίκη, να αναψηλευστεί η δίκη και να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα δίκαιας δίκης του ακτιβιστή από την Κυριαζία. Κύριο κύριος Χάουιτ, έχετε να προσθέσετε κάτι? Θα ήθελα να σας πω ότι σας ευχαριστούμε θερμά για τις ανακοινώσεις. Ήταν πολύ ενημερωτικές και πολύ χρήσιμες και είναι σημαντικό για τα πρακτικά να αναφερθεί αυτό συμφωνώ απόλυτα και υποστηρίζω όλες τις συστάσεις σας. Καταρχήν, στις 6 Δεκεμβρίου είχα ζητήσει να προσθεθεί ένα επιπλέον σημείο. Βέβαια δεν, δεν τα κανονίζουμε όλα αυτά στο Προεδρείο και τελικά στις 6 Δεκεμβρίου θα έχουμε μια σημαντική συνεδρία στις Βρυξέλλες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και θα ήθελα στην συνεδρίαση 6 Δεκεμβρίου να προβλέψουμε ένα λίγο χρόνο. Όντω έχουμε πάρα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα φροντίσουμε συνεδρίαση 6 Δεκεμβρίου να συμπεριλάβουμε και τη δική σα πρόταση. Πάντω, με την κυρία Σάρκε, την κυρία Μαρίτσια Σάρκε, καταθέσαμε χθε δύο ερωτήσει προ το Συμβούλιο και την Επιτροπή σε ό,τι αφορά τι προθέσει του για, τα, για τις διεθνείς προδιαγραφές τηλεπικοινωνιών και την εξαγωγή τεχνολογιών παρακολούθησης, ιδιαίτερα όταν τέτοιου είδους τεχνολογίες παρακολούθησης και υποκλοπής χρησιμοποιούνται για να ελεγχθούν οι κινήσεις ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό να συνεργαστούμε με τις επιχειρήσεις για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των ακτιβιστών και να μην γίνεται κατάχρηση τέτοιων τεχνολογιών. Επίσης, τον Ιούνιο ε, ακούσαμε την ομολογία της ε, Nokia και της Siemens γιατί οι εταιρείε αυτές αναγνώρισαν στην σχετική ακρόση που είχαμε για το ίντερνετ ότι δεν είχαν αντιληφθεί σωστά την κατάσταση στο Ιράν και έκαναν λάθη εξαιτία αυτής της παρανόησης. Τώρα έχουν εκφράσει την επιθυμία να συνεργαστούν για την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Βέβαια, οι ανταγωνιστές τους από την Ευρώπη και την Κίνα δυστυχώς ε, δεν έχουν τέτοιου ενδιασμούς και δυστυχώς ίσω εφαρμόσουν εμπορικέ πρακτικές που θα οδηγήσουν σε καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Και τώρα ας περάσουμε στο κυρίως θέμα της πρωινή μα συζήτηση. Στις 10 Οκτωβρίου έχουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινή Και από τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει πρωταρχικό τη στόχο και προτεραιότητα την ολοσχερή κατάργηση της θανατικής ποινής στον κόσμο είναι πολύ επίκαιρο να διοργανώσουμε και εμείς μια δημόσια κρόαση για το θέμα αυτό και έχουμε και επιφανείς προσκεκλημένους για παράδειγμα τον κύριο Κλάιβ Στάφορτ Σμιθ δικηγόρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και διευθυντή της Reprieve, μιας Βρετανικής ε, οργάνωσης σας καλωσορίζουμε θερμά κύριε Στάφορντ γιατί ξέρουμε ότι εργάζεστε πολύ σκληρά για να προωθήσετε το μορατόριο της θανατικής ποινής, ιδιαίτερα εις βάρος ε, Ευρωπαίων Υπηκών. Έχουμε μαζί μας και τον κύριο ε, Σόουζα που είναι ο νομικός σύμβουλος της Μεξικανικής Πρεσβείας. Γνωρίζουμε κύριε Σόουζα ότι έχουμε μια μεγάλη, ένα μεγάλο αριθμό δυστυχώς μεξικανών υπηκών που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναμένουν εκτέλεση. Έχουμε και τον κύριο Ραφαέλ Σενουί Χαζάν, εκτελεστικό διευθυντή της Παγκόσμιας Συμμαχίας κατά της θανατικής ποινής. Καλώς ήρθατε και βλέπω με χαρά τον κύριο Μάικλ Τίλεμανς, τον πρόεδρο της ΚΟΧΟΜ, εκ μέρους της Βελικής Προεδρίας. Και φυσικά θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά και την κυρία Βερονίκ Αρνό, Διευθύντρια των Πολυμερών Σχέσεων και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Αρμόδια Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων της ευρωπαϊκή Επιτροπής. Εν είδη αγωγή, ήθελα να σα υπενθυμίσω την ε, στεναρή προσήλωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για την κατάργηση τη θανατική ποινή. Με βάση τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μα, γνωρίζουμε ότι 154 χώρε και εδάφη που σε διαφορετικού βαθμού αποφάσισαν να αποκηρύξουν τη θανατική ποινή. Και αν δεν κάνω λάθο, η κυρία Λόχ Μπίλερ επισήμανε στην συζήτηση τη περασμένη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι όντω αυτό συνιστά επιτυχία, αλλά δεν έχουμε υλοποιήσει ακόμη τον τελικό μας στόχο, γιατί οι χώρες που εφαρμόζουν την θανατική ποινή διεθνώ είναι 43 πια, αρχικά ήταν 48. Ε, το 2008 μάλλον οι χώρες αυτές ήταν 48. Βλέπετε υπάρχει μια μείωση των χωρών που μένουν στη θανατική ποινή. Το 2009 ο αριθμός των χωρών που εφάρμοζαν τη θανατική ποινή ήταν 18, σημαντική μείωση δηλαδή του αριθμού των χωρών και η σταδιακή εγκατάλειψη της θανατικής ποινής είναι προφανής ε, γιατί ακόμη και χώρες που προβλέπουν στο ποινικό του σύστημα τη θανατική ποινή ως την εσχάτη των ποινών δεν την ε, εφαρμόζουν παρόλα αυτά. Και με βάση τις στατιστικές του 2009 είχαμε 5.000 και εκτελέσεις λίγες λιγότερες από τις 5.700 το 2008. Υπήρξε μια σταδιακή μείωση γιατί το 2007 είχαμε έναν ακόμη μεγαλύτερο αριθμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναλαμβάνω, είναι αναφαδόν κατά της θανατικής ποινής. Η κατάργηση της θανατικής ποινής διεθνώς αποτελεί από τους πρωταρχικούς στόχους τη πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί που υπάρχει ακόμη και ισχύει η θανατική ποινή, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλή για τη σταδιακό περιορισμό της ε, επιβολής, σεβασμό των ελάχιστων ε, προδιαγραφών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατά πάσα πιθανότητα το θέμα της θανατικής ποινής θα ε, απασχολήσει και πάλι την Γενική Συνέλευση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τι επόμενε εβδομάδε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε και σχετικό ψήφισμα εν ώψη τη Παγκόσμια ημέρα κατά τη θανατική ποινή στι 7 Οκτωβρίου. Ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προέβηκε σε δήλωση στι 8 Οκτωβρίου και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης συνέταξαν κοινή διακήρυξη την ίδια μέρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όλα αυτά τα έγγραφα σας έχουν διανεμηθεί και τέλος πριν περάσουμε στην ακρόαση με τους επιφανείς μας προσκεκλημένους θα ήθελα να τονίσω το έργο του δόκτωρα Clive Stafford Smith. Και μάλιστα μετά το πέρα συνεδρίες στη μία οργανώνουμε συνέντευξη τύπου στην οποία είστε προσκεκλημένοι όλοι. Ο δόκτωρας Clive Στάφορτ Σμιθ θα μας παρουσιάσει μια μελέτη για τους Ευρωπαίους πολίτες που ονομένουν εκτέλεση τη θανατικής του ποινή στον κόσμο. Παρακαλώ να μην ξεπεράσετε τα δεκάλεπτα στην παρουσίασή σας για να προλάβουμε να έχουμε και δεύτερο γύρο με απαντήσει. Δόκτωρα Στάφορτ Σμιθ, έχετε το λόγο. Ah, there we go. Even as a lawyer, ε, παρότι είμαι δικηγόρος θα προσπαθήσω να μην μιλήσω πάνω από 10 λεπτά. Είναι μεγάλη τιμή που με προσκαλέσατε σήμερα. Είμαι Αμερικανός και ε, ε, Βρετανός. Είμαι λίγο σχιζοφρενής. Θα μιλήσω όμως ως Αμερικανός για να μιλήσω από εξ ονόματος κάποιας χώρας που διατηρεί την θανατική πίνη. Σας ευχαριστώ όλους για τη δουλειά που έχετε κάνει. Χθες το βράδυ πήρα ένα γράμμα από μία συνάδελφο στην Καλιφόρνια και μου είπε να σας το παραδώσω ο Μάλκο Μένεν ε, που εκπροσωπεί ε, πάνω από 700 μελοθάνατους ε, στη ΣΥΠΑ και θα ήθελε να τονίσει και εγώ θα ήθελα να το πω αυτό ότι είμαστε ευγνώμονες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για, την, για τα όσα έχετε καταφέρει κατά της θανατικής ποινής δηλαδή θα μας δίνετε μέχρι να επιστρέψουμε επιτέλους στον πολιτισμό κι εμείς Σα ε, σας ευχαριστούμε. Ε, μιλώ με την ιδιότητα ε, του Διευθυντή του, Οργανισμού Reprieve που λαμβάνει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ύπατη Ερμοσία του ΟΗΕ αλλά δεν περιοριζόμαστε σε αυτό και δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι μας χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο αλλά ήθελα να σας πω ότι για μας και για όσους ανά τον κόσμο ε, ε, περασπίζονται ε, την κατάργηση της θανατικής ποινής. Εκπροσωπούμε πάνω από 300 φυλακισμένους που περιμένουν εκτέλεση της θανατικής ποινής και έχουμε άμεση γνώση του τι θα μπορούσε να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί πράγμα μιλάμε, αυτό που είπατε, συνεργασία, τίποτα δεν υπάρχει από αυτά που να ζητάμε που πρόκειται να επιβάλλει οτιδήποτε στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν σας υποδείξουμε εμεί ποιο δρόμο θα ακολουθήσετε. Θέλουμε να συνεργαστούμε με όλες τις κυβερνήσει, ούτως ώστε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο να παρεμβαίνουμε, αν κατά περίπτωση. Ο κύριο Σίζερ εκπροσωπείται εδώ πέρα το Μεξικό με τον πρέσβη ε, Σίζερ και είναι ένα λαμπρό παράδειγμα γιατί... Ε, η Αμερικανική κυβέρνηση έχει υποστηρίξει αυτούς τους ε, κρατούμενους ε, στο Μεξικό που αντιμετωπίζουν την θανατική ποινή και έχουμε μπλακεί άμεσα σε αυτό το, σε αυτή, στις μεξικανικές περιπτώσεις. Και Εάν ε, υπάρχει τέτοια δραστηριότητα, υπάρχουν πενταπλάσιε δυνατότητες να αποφύγουμε τη χρήση τη θανατική ποινή. και νομίζω ότι για τέτοιου είδου συνεργασίε θα πρέπει να μιλάμε. Τώρα ποιο είναι το όφελο στο να έχουμε μια παρέμβαση από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποιου κράτους μέλου για του υπηκόου του. Μην υποτιμάτε τη σημασία ενό τέτοιου εγχειρήματο. Ε, το 1995 συναντήθηκαμε με την Ίγμεν και εμεί ήμασταν στο Κέμπριτζ μαζί ε, ε, και τι είχε συμβεί ε, τότε, ήταν να παρέμβει η Βρετανική κυβέρνηση και συζήτησα με την, το, το δικηγόρο του και μου είπε ότι αν η Βρετανική κυβέρνηση είχε απλώς ζητήσει η Ικτό, η Νίκη ε, θα ήταν ακόμη ε, ζωντανή σήμερα. Ε, έχει είχε αλλάξει στάση η Βρετανική κυβέρνηση και παρεμβαίνει πολλές φορές για να υπερασπιστεί Βρετανούς υπηκόους που αντιμετωπίζουν θανατική ποινή στη ΣΥΠΑ ή σε κάποια άλλη χώρα. Ο Νίλ Ρέβερ, μια άλλη περίπτωση πριν από κάποιους μήνες ε, που ε, ε, αντιμετώπιζε θανατική ποινή, αλλά τελικά εξέφυγε από αυτό τον κίνδυνο χάρη στην παρέμβασή της βρετανική κυβέρνηση και νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει από πλευράς διαφόρων κυβερνήσεων ακόμη και όταν κάποιος δεν είναι υπήκος μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά διαμείνει και ο Χαν Σκίνερ εσχάτως έφτασε στα 35 λεπτά πριν την εκτέλεσή του και χάρισε στον πρόεδρο Σαρκοζή σώθηκε, ήταν απλώς παντρεμένος με μια γαλίδα υπήκο και ε, χάρισε στην παρέμβαση του πρόεδρου Σαρκοζή, ε, γλίτωσε ενώ είχε φτάσει στα 35 ε, λεπτά από την εκτέλεση. Άλλες περιπτώσεις είναι 58 δεύτερα πριν την εκτέλεση. Περί αυτού πρόκειται σήμερα. Πώς, με ποιο τρόπο μπορούμε να καταστήσουμε όλο και πιο αποτελεσματικέ παρεμβάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι πρέπει να κάνουμε, πρώτα απ' όλα να εντοπίσουμε ποιοι είναι οι μελοθάνατοι, ποιοι αντιμετωπίζουν ε, ε, την θανατική ποινή σε ε, άλλε χώρε. Στη ΣΥΠΑ κάνουμε μία έρευνα για όλους τους 3.263 που αντιμετωπίζουν θανατική ποινή για να εντοπίσουμε ποιοι είναι Ευρωπαίοι και ποιοι είναι οι υπήκοοι άλλων χωρών. Ο Μάλκον Ρένελ που σας στέλνει αυτή την επιστολή από την Καλιφόρνια αναφέρει ότι τουλάχιστον 50 υπήκοοι ε, ε, υπάρχουν σε άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν θανατική ποινή και 150 που έχουν σχέσεις ε, γάμο ή οτιδήποτε άλλο με υπηκό των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τον κόσμο και ε, το ΙΠΑ είναι ένα μικρό κομμάτι του προβλήματος. Ε, στο Πακιστάν, παραδείγματος χάρη, 7.500 περιμένουν την εκτέλεσή τους ε, και εκπροσωπούμε κάποιους Βρετανούς επικούς εκεί στο Πακιστάν και κανείς δεν ξέρει τίποτα για αυτούς, από όσους ξέρω εγώ. Γι' αυτό σας λέω, το σημαντικό είναι να εντοπίσουμε τους επικούς ε, κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που ε, αντιμετωπίζουν αυτή την απειλή σε άλλες χώρες. Και επίσης μας βοηθάει πάρα πολύ η συνεργασία μαζί σας σε αυτή τη διαδικασία εντοπισμού. Τώρα έχουμε ένα νόμιμα δικαίωμα να παρέμβουμε και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αναφέρει ότι βασικό λειτουργήμα ε, των δημοσίων υπαλλήλων των ΗΠΑ είναι να επικουρούν τους υπηκούς ε, των χωρών αυτών. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να συγκλίνουν όλε οι προσπάθειε ε, και μεταξύ των οποίων και του ΟΗΕ για την κατάργηση τη θανατική Ποινή, ούτως ώστε να γίνονται αποτελεσματικέ παρεμβάσει. Οι Μεξικανοί θα μα το πούν πώ ακριβώ έχουν κινηθεί, γιατί ε, είχαν λαμπρά αποτελέσματα. Ε, και η οργάνωσή μα, ΡΕΠΡΙΒ, έχει συνεργαστεί με το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και με άλλε χώρε. και θα ήθελα να τονίσω ότι πριν από δύο εβδομάδε ο διαμεσολαβητή μα, ε, στην ε, ο διαμεσολαβητή στην Ουκρανία μα βοήθησε πάρα πολύ γιατί τάχιστα μα έδωσε τι απαιτούμενε πληροφορίε για να βοηθήσουμε του δικού υπηκούς που αντιμετωπίζαν θανατική ποινή στην Βιρτζίνια. Πώ μπορούμε να συγκροτήσουμε αυτό τον συνασπισμό με τι κυβερνήσει, μη κυβερνητικέ οργανώσει, Ευρωπαϊκέ χώρε και σε χώρε ανά τον κόσμο, ώστε να εντοπίσουμε, να οριοθετήσουμε συγκεκριμένα το πρόβλημα και να βοηθήσουμε αυτού ε, του ε, υπηκόου αυτών των χωρών. Και δεν θέλουμε να βοηθήσουμε μόνο υπηκόου ευρωπαϊκών χωρών. Ε, Απλώ νομιμοποιείται περισσότερο η παρέμβασή μα, αλλά ταυτόχρονα όμω έτσι βοηθάμε και πολλού άλλου που αντιμετωπίζουν τη θανατική ποινή ανά τον κόσμο. Στην Ιεμένη είχα ενδιαφέρουσε συζητήσει. Ε, με διάφορα στελέχη που αναγνώρισαν πόσο σημαντικό είναι το θέμα, αλλά νόμιζαν ότι έρχομαι από τον Άρη που ε, αντιτάσσομαι στην θανατική ποινή και εκπροσωπούσαμε κάποιους που αντιμετωπίζουν τη θανατική ποινή στην Ιεμένη και υποστηρίζοντας αυτούς ε, βοηθούμε και τους υπόλοιπους κρατουμένους σε αυτή, σε αυτή τη χώρα. Πολλέ φορέ εκπροσωπούνται οι φυλακισμένοι κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν καταλαβαίνουν όμω πλήρω το πρόβλημα. η εκπροσωποί του θα μπορέσουμε να το ξανασυζητήσουμε και μέχρι τότε θα περιμένω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα σα ευχαριστώ, ήσασταν πάρα πολύ σύντομο. Ναι, 8 λεπτά έκανα μόνο. Κοίταξε και το ρολόι. Στη Αμερικάνικα διαστήρια σου δίνουν μία ξυλιά αν ξεπεράσει το χρόνο. Γι' αυτό είμαι μαθημένο. Ωραία. Ο κύριος Σούζα τώρα θα πρέπει να πάρει το ε, λόγο για να μας πει πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος της μαξικανικής κυβέρνησης στην εξαρτή αυτή. Παρακαλώ κύριε Σούζα, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για τρία λεπτά περίπου. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για την ακρόασή σας αυτή στην ακρόαση. Ε, έχω έτσι δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψη όσον αφορά τις κύριες πράξεις ε, μεξικανικής κυβέρνηση και του Υπουργείου Εξωτερικών για προστασία μεξικανών υπηκών στο εξωτερικό. Ιδίως πρόκειται για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκείνων που απειλούνται από την θενατική πηγή και πρόκειται για το θέμα της ε, ε, νομικής υποστήριξης, προσπάθειες μέσω των διπλωματικών εκπροσω... και κλπ. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα για την ε, εξατία μας αυτά σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο. Και μάλιστα κάναμε και ένα διάβημα στο Αμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζητώντα σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του συμφώνου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εφαρμογή τους ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επιβολή θανατικής ποινής σε αλλοδαπούς υπηκόους. Γιατί μερικές φορές χρειάστηκε να προσφύγουμε στη βοήθεια των προξενικών αρχών και μάλιστα αυτό το προηγούμενο ήταν από τις σημαντικότερες βάσεις που χρησιμοποιήθηκε αργότερα και σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο ως σημείο αναφορά σε ό,τι αφορά ε, τις ε, αποφάσεις ενός πολύ σημαντικού οργάνου. Το διαμερικανικό ε, Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, είχε συνεργασία με το, τη Μεξικανική κυβέρνηση προκειμένου να, παρέσ, να παράσχει ειδική δικαστική αρρωγή σε Μεξικανούς επικόους που αντιμετώπιζαν θανατική καταδίκηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα το πρόγραμμα αυτό συνεχίστηκε και από το 2001 εφαρμόζεται όλο και περισσότερο και μάλιστα καλύπτει όχι όσους έχουν καταδικαστεί σε θάνατο αλλά και όσους ε, έχοντας διαπράξει έγκλημα ε, θα αντιμετώπιζαν ε, πιθανότητα καταδίκη σε θάνατο. Οπότε το πρόγραμμα αυτό ήταν πολύ σημαντικό και βασικός του στόχος ήταν να πετύχει αναστολή της καταδίκης η ακύρωση της θανατικής ποινής χάρη σε ένδικα μέσα και δικαστικής αρρωγής, ιδιαίτερα της, των συνηγόρων των καταδικασμένων. Γιατί το Αμερικανικό Δίκαιο περιλαμβάνει πολλές δικονομικές εγγύσεις που θα πρέπει να πληρούνται από τους συνηγόρους, ιδιαίτερα σε, σε υποθέσεις θανατικής ποινής και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τη ζωή των δικηγόρων σε τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης έχουμε πολλές φορές σύγκρουση του Αμερικανικού Δικαίου με το Διεθνές Δίκαιο και ήταν πολύ δύσκολες πολλές φορές να πετύχουμε ακύρωση ή αναψηλάφιση μιας τέτοιας υπόθεσης. Βέβαια μερικές φορές έχουμε ακρόαση μαρτύρων στο Μεξικό ή διάφορες εμπειρογνωμοσύνες ή ψυχολογική ε, εξέταση, όλοι αυτοί οι λόγοι μπορούν να συμβάλλουν στην ακύρωση ή αναβολή της θανατικής ποινής. Επαναλαμβάνω, το πρόγραμμα του 2001 εξελίσσεται συνεχώς και προσπαθούμε να προσδιορίσουμε ποια στιγμή ένας ειδικευμένος δικηγόρος μπορεί να επέμβει και ποια στιγμή ε, περιπτώσεις ε, εγκλημάτων μπορούν να οδηγήσουν σε επιβολή θανατικής ποινής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να βρούμε αυτή την κατάλληλη στιγμή και αυτό και χρειάζεται κατάρτιση και των δικηγόρων και εγώ μάλιστα ήμουν σε μια παραμεθόρια ζώνη του Τέξας και πολλές φορές είναι κρίσιμες οι πρώτες ώρες ε, της κράτησης για να αποφευχθεί αργότερα τέτοιου είδους ε, θανατική καταδίκη. Έχουν γίνει σημαντικές ε, προσπάθειες κατάρτισης των προξενικών αρχών. Έχουμε το σημαντικότερο προξενικό δίκτυο που έχει μία χώρα σε άλλη. Έχουμε 50 προξενία στις Ηνωμένε Πολιτείες. Η μεγαλύτερη προξενική παρουσία ξένης χώρας στις Ηνωμένε Πολιτείες. Και μας ενδιαφέρει φυσικά η προστασία των Μεξικανών επικών στα πλαίσια αυτής αυτού του δικτύου. Έχουμε επίση μια ένωση δικηγόρων που δικεύονται σε ε, υπεράσπιση καταδικασέντων σε θανατική ποινή και επίση ε, ένα δίκτυο εμπειρογνώμων ε, για θέματα ψυχιατρικά, νευροψυχιατρικά κτλ. Όπως ε, μας είπε ο Δ. Στάφορτ, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για την μελέτη του, χάρη στο πρόγραμμα αυτό έχουν, έχει μειωθεί η εκτέλεση των θανατικών ποινών από τις, από τις 545 περιπτώσεις 9 μόνο καταδικάστηκαν σε θάνατο και αυτή τη στιγμή, χάρη στην εφαρμογή του προγράμματος και η επέμβαση του προγράμματος μέχρι στιγμής για την αναστολή των θανατικών ποινών είναι το 1% και θα ήθελα να εκφράσω την αναγνώρισή μου προς το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έργο της. Πρόσφατα είχαμε την επιστολή της ε, κυρίας Άστον στην Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην κυρία Κλίντον και επίσης πολλές αλληλέγγυες ε, πρωτοβουλίες και διαβήματα από το Συμβούλιο της Ευρώπης, από ευρωβουλευτές, αλλά και το... η σημαντική προσήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το στόχο της ε, κατάργησης θανατικής ποινής. Θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά όλες τις ε, οργανώσεις που δίνουν μάχη, αλλά και τους δικηγόρους που υπερασπίζουν καταδικασέντες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση σε αυτή και τις προφήσεις που μας δώσετε για τις μεσχανικές δραστηριότητες και την ενδυνάμωση της ε, συνεργασίας. Θα ήθελα τώρα να καλέσω τον κύριο Ραφαέλ Σινουιλιαζάν, εκτελεστικό διευθυντή του Διεθνού Συνασπισμού κατά της θανητικής ποινής. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, είμαι γενικός ε, διευθύντης της GPM, ε, διεθνούς ε, συναπισμού κατά τη θανατικής ποινής, ε, οργανώσεις που συνενώνει πάνω από 100 οργανώσεις ανά τον κόσμο. Η γραμματεία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μου ζήτησε να κάνω μια γενική παρουσίαση της κατάστασης κατά της θανατικής ποινής. Προχθές ήταν η Διεθνή Σημέρα κατά ποινή. Αυτή είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να εξτάσει κανένας και να δει τι συμβαίνει ακριβώς. Η πρώτη παρατήρηση είναι μια σημαντική πρόοδο υπέρ τη κατάργηση. Σήμερα 139 χώρε έχουν καταργήσει θανατική ποινή, είτε de jure είτε de facto. Οι ε, ορισμένε άλλες χώρε εξακολουθούν να διατηρούν αυτή την ποινή. Το 2009 μόνο 18 χώρες ε, εκτέλεσαν ε, τις θανατικές πηγές. Ε, υπάρχει γενικά ένα δημοσιακό κίνημα κατά της καταρρύξης. Το 1981 35 χώρες είχαν καταργήσει θανατική ποινή. Ενώ σήμερα τα δύο τρίτα όλων των χωρών από τον κόσμο έχουν καταργήσει θανατική ποινή, είτε στην πράξη είτε ε, δια τα τελευταία παραδείγματα το μπορούν και η Ρουάντα το 2008, το Τόγκο το 2009 ή ε, τη πολιτεία του Νέου Μεξικού το 2009 επίσης. Παρ' όλα αυτά η κατάσταση είναι δύσκολη σε ορισμένε περιοχές του κόσμου. Στην Κίνα παραδείγματο χάρη. Το αναφέρατε κι εσείς πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτή τη χώρα για το θέμα της αντικής ποινής υπάρχει πραγματικό πρόβλημα διαφάνειας όσον αφορά την, ε, το πραγματικό ρυθμό εκτελέσεων. Εκτιμούμε ότι υπάρχουν 6.000 εκτελέσεις ανά έτος. Αλλά για το 2009, παραδείγματο χάρη, έχουμε μονάχα επίσημα αναγνωρισμένε 714 εκτελέσεις. Ο δεύτερο μεγάλος ε, τομέας είναι η Ανατολή. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στι Ισλαμικές χώρε που, όπου, που διάπονται από τον νόμο τη Σαρία. Στο Ιράν ιδίω. με πάνω από 388 εκτελέσει το 2009. Και ιδίω μετά τι εκλογέ του Ιουνίου του 2009. <clears throat> μετά έχουμε τη ΣΥΠΑ που ανέφερε και ο Κλίβ στην παρουσίασή του. Εννέα πολιτείες εκτέλεσαν θανατικέ πηγές ε, το 2009, ε, θανατώντας 52 άτομα. 2.380 άτομα βρίσκονται αυτή τη στιγμή εν αναμόνη της εκτέλεσης θανατική του Βλέπουμε μείωση λοιπόν των εκτελέσεων και στη χώρα αυτή. Η ΕΠΑ είναι μία από τις σπάνιες δημοκρατίες, 7 στο σύνολό που καταδικάζουν και εκτελούν ανθρώπου ανά τον κόσμο. Γενικά η είναι ακριβώς ένα αντιπαράδειγμα που πολλές χώρες χρησιμοποιούν για να δικαιολογήσουν την δική τους ε, θανατική ποινή. Δύο λόγια όσον αφορά τη λειτουργία του... Τα, τα θύματα στο Ιράν μπορούν να είναι γυναίκες, όμως φιλόφιλοι νέοι, παραδείγματο χάρη ανήλικοι δηλαδή, στο Ιράν, στη Δαούδια Βόρεια στη Γερμανία, 59 ανήλικοι εκτελέστηκαν το 2009. Μπορεί επίσης να είναι άτομα με ε, πνευματικές καθυστερήσεις. Πριν από δύο ε, εβδομάδες εκτελέστηκε ο Ζαρουής στη Βιργινία με ένα δίκτυο νοημοσύνης μεταξύ του 70 και του 72 μπορούν επίσης να ανοίξουν σε μειονότητες εθνοτικέ, ή, ή όπω ε, θρησκευτικές, όπως παραδείγματο χάρη στις ε, χώρες του κόλπου του Περσικού κόλπου ή μπορούν να είναι θύματα πολιτικής καταστολής όπως το Ιράν στην Κίνα και σε άλλες τόσες χώρες. Εν κατακλείδη θα ήθελα να τονίσω τις στάσεις για το μέλλον και τα νέα μέτωπα μάχης. Γεωγραφικά βέβαια η Μέση Ανατολή, η Ασία και η ΙΠΑ εξακολουθούν να παραμένουν οι προτεραιότητε μας. Ανησυχούμε όμως για την κατάσταση στην Κεντρική Αμερική, στη Γουατεμάλα ιδίω και στην Ικαράγουα, όπου συνεχίζονται οι συζητήσεις για την επανεισαγωγή της αρνητικής ποινής. Θεματικά τώρα. Το εμπόριο ναρκωτικών είναι ένα προβληματικό θέμα για τα τελευταία, τα δύο χρόνια και για το μέλλον. Πολλές χώρες έχουν κατά νου να επανεισαχθεί η θανατική ποινή για αυτούς τους λόγους. Παραδείγματος κάνει και τη Νότια Αμερική. Πολλές από τις καταδίκες γίνονται για αυτούς τους λόγους και επίσης στην Κίνα και στην Ασία. Επίσης το επιχείρημα της τρομοκρατίας είναι σημαντικό και θα μας απασχολεί στα επόμενα δύο έτη. Επίσης ένα σημαντικό θέμα είναι ο σχετισμός μεταξύ του Ισλάμ και της Ανατικής ποινής, ε, μεταξύ του νόμου της Σαρία και της Ανατικής ποινής. Ε, αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουμε σημαντικά υπόψη για το μέλλον. Αυτό που μας κάνει ελπίζουμε είναι το μορατόριο στη Μογγολία πρόσφατα, τα μελλοντικά ενδεχομένω ε, μέτρα που θα αναλάβει η Λευκορωσία. Τα θετικά μηνύματα από την Αφρική, το Μάλι, το Γκαμπούν και άλλες χώρες και στην Ασία μια πολιτική βούληση να μην εκτελούνται οι ε, τα άτομα αυτά στην ε, Μογγολία παραδείγματο χάρη. Η κοινωνία των πολιτών, οι κυβερνήσει και οι διεθνείς οργανώσεις έχουν ασκήσει πίεση και συνεργάζονται παραδείγματο χάρη μέσα στα πλαίσια του Διεθνού Συνεδρίου κατά θανατικής πηγής παραγωγών ECPM ή την πρόσφατη δημιουργία της Διεθνής ε, Επιτροπής με πρωτοβουλία της Ισπανικής Κυβέρνησης που ξεκίνησε στη Μαδρίτη την περασμένη εβδομάδα. Οπωσδήποτε, ο δρόμος προς την ε, κατάρριση της ελληνικής πηγής δεν πρόκειται να εστρεφεί. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε και για τις ελπίδες που μας δώσατε για αυτές τις χώρες που τώρα προς... Ε, προσεχώς θα καταργήσουν την θανατική πηγή και ιδίως αναφερθήκατε και στη Λευκορωσία, μια πολύ περίπτωση γιατί μια από τι χώρε τη ε, ανατολική εταιρική σχέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Θα ήθελα να στραπώ τώρα στα ευρωπαϊκά όργανα. Έχουμε τον κύριο Τίλεμαν, πρόεδρο τη ΚΟΧΟΜ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας καλέσω για την πρόσκλησή σας και να χαιρετήσω επί τη ευκαιρία όλα τα μέλη της Υποεπιτροπής σας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σήμερα, Πρόεδρε, θα ήθελα να εστιάσω την ε, παρέμβασή μου στο σχέδιο ψηφίσματος που ευρημάζεται ε, στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και για να μπορέσω να είμαι κατανοητό στο ε, Ηνωμένα Έθνη θα μιλήσω αγγλικά. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω όταν προετοιμάζαμε το δε, ε, πρόγραμμα 18 μηνών του τρίου της ε, Προεδρίας, ε, των Προεδρεών που τελειώνουμε τη Βελική Προεδρία, το θέμα της ανθρώπινης, της χρονικής πηγής ήταν το πιο σημαντικό και είχαμε συμφωνήσει ότι η κατάρριξη της θανατικής ποινής θα παρέμενε στη μεσαία διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα διεθνή θέματα. Και γι' αυτό το Βέλγιο αποφάσισε ένα από τα εργαστήρια του Φόρουμ ε, ε, για να, ασχοληθεί με, τα, με την Αθλαντική Πηγή στις 13 Ιουλίου και εξετάστηκε το θέμα των μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα στα πλαίσια συνθήκης του Λισαβόνα. Αυτό το εργαστήριο που αφορούσε συγκεκριμένα την ειδική ποινή και πώς η συνθήκη του Λισαβόνα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγές. Και εκεί η κοινωνία των πολιτών υπέβαλε μια σειρά ε, συστάσεων. Δεν θα επισέλθω σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά θα ήθελα να τονίσω τους κύριους προσανατολισμούς. Καταρχήν συνοχή και συνέπεια. Δεύτερον, συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Τρίτον, παιδεία και ε, δημιουργία ε, κινητοποίησης αποτελεσματικότητα επίσης, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και να αξιολογήσουμε πού μπορούμε κάτι να βελτιώσουμε στην συμπεριφορά μας. Δύο από αυτές τις συγκεκριμένες ε, συστάσεις θα ήθελα να τις τονίσω ιδιαίτερα. Πρώτον, Κατήχαμε στο στα συμπέρασμα σε αυτό το φόρουμ ότι η οργάνωση σεμιναρίων στα Εθνικά Κοινοβούλια και η οργάνωση ενός δικτύου βουλευτών για την κατάρριξη της στρατηγικής ποινής ήταν κάτι που ε, έπρεπε να τύχει υποστήριξης. Δεύτερον, να προωθήσουμε την διαφάνεια όσον αφορά τις χώρες, τις χώρες στις οποίες εξακολουθεί να υπάρχει θενατική πίνη ζητώντας πληροφορίες για τις εκτελέσεις να αποστέλουν στην ΕΠΑ το εκπρόσωπο, την κυρία Άστον. Ο λόγος για τον οποίο τονίζω τελείως αυτές τις τάσεις είναι γιατί θα ήθελα να σας πω ότι εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει στη δημιουργία του δικτύου αυτού με άλλους εταίρους ε, εθνικού ή περιφερειακού χαρακτήρα. Στρεφόμενος τώρα στο θέμα των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει μια σειρά εκθέσεων που υπευλήθησαν από τα διάφορα σώματα των ε, Ηνωμένων Εθνών, ιδίως από το Γενικό Γραμματέα, πρόσφατα. Και όπως ακούσαμε σήμερα, από τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών πραγματικά υπάρχει μια τάση προς μορατόριο ή και κατάργηση της θανατικής ποινής. Όλα αυτά, αυτές οι εκθέσεις τονίζουν το γεγονός ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τις χώρες αυτές οι οποίες εξακολουθούν να ε, διατηρούν τη θανατική ποινή να είναι πιο διαφανείς και μια από τις ανησυχίε του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ ήταν ακριβώς η έλλειψη βασίμων στοιχείων για τις εκτελέσεις. Ένας από τους ομιλητές μόλις τώρα τόνισε ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Και αναφέρθηκε σε μια συγκεκριμένη χώρα με στοιχεία αριθμητικά. Τώρα τι θα κάνουμε στην ίδια Συνέλευση των Ηνωμένων τώρα εμείς και όταν λέω εμείς δεν εννοώ μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μια τεράστια ομάδα χωρών που έχουν τις ίδιες απόψεις με μας θα εισαγάγουμε, θα υποβάλουμε ένα ψήφισμα στην, ε, στην αρμόδια επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης και μετά στην ίδια τη Γενική Συνέλευση. Αυτό που είναι σημαντικό για μας, και είναι η κύρια μας προτεραιότητα, είναι το ψήφισμα αυτό να επιβεβαιώσει και να τονίσει αυτή την τάση που όσο πάει και αυξάνεται για την υποστήριξη του μαρατόριου για θανατική ποινή. υπάρχουν παρόμοιες, ε, παρόμοια ψηφίσματα το 2007-2008, αλλά τώρα θα έχουμε πιο έντονα στοιχεία και απαιτήσει. Την περασμένη φορά μάλιστα τα, τα ψηφίσματα αυτά υποστηρίξαν από 89 κράτη-μέλη της ε, συνέλευσης και 105 ε, χώρες υπερψήφισαν. δεν Θα τονίσω ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονη υποστήριξη του ψηφίσματος. Αποφασίσαμε να έχουμε στη Νέα Υόρκη μια task force που να αποτελείται από κύριους συμμετέχοντα από όλες τις περιφερειακές ομάδες Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες περιφερειακές ομάδες για να διευκολύνουμε τη διαδικασία και να διευκολύνουμε την εργασία εκείνων που υποστηρίζουν το ψήφισμα να μπορούν να το υποβάλουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλος του Task Force φυσικά, αλλά επίσης η Αγγόλα, η Αργεντινή, το Μπουρούντι, η Χιλή, το Ανατολικό Τιμόρ μεταξύ άλλων. Τώρα, όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Νέα Υόρκη. Καταρχήν έχει συμφωνηθεί ένα κείμενο από τους συνυποβάλλοντες. Πολύ γλυκόρα προχώρησε η διαδικασία. Και αν όλα πάνε όπως ε, είναι τα σχέδιά μας, το ψήφισμα θα υποβληθεί την επόμενη εβδομάδα στα Ηνωμένα Έθνη. Δεν θέλω επίσης να τονίσω ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτές οι χώρες μέλη του ΟΗΕ που υποστηρίζουν αυτό το ψήφισμα θα ξεκινήσουν με μεγάλη εκστρατεία για να προχωρήσει το ψήφισμα. Θα υπάρχει πολύ lobbying δηλαδή για την υποστήριξη του ψηφίσματος που υποβάλλεται. Δύο τελευταία σημεία. Καταρχήν, από τι επαφέ με ορισμένε χώρε που διατηρούν την θανατική ποινή που είναι πιο πλησίων ημών από ό,τι άλλε, ότι θα, δούνε με, θα ακούσουμε βίκο ε, το ψήφισμα αυτό. Καλό είναι αυτό να το ξέρουμε λοιπόν. Ακόμα δηλαδή και εκείνα τα κράτη-μέλη του ΗΠΑ που δεν μπορούν να μας υποστηρίξουν, καμιά φορά συνεργάζονται μαζί μας. Το δεύτερο είναι ότι εκτός από το ψήφισμα είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στις διμερείς επαφές η Ευρωπαϊκή Ένωση συστηματικά θέτει το θέμα σαν ειδικής ποινής σε χώρες εταίρους, στους διαλόγους, στις διαβουλεύσεις. Και θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι με μια σειρά χωρών, με όλες τις χώρες κατά βάση, προσπαθούμε να αναπτύξουμε ομάδες πιέσεις με διακριτικές ή λιγότερο διακριτικές πράξεις για να μπορέσουμε να τους κινήσουμε προς την ε, πολιτική αυτή. Μπορεί κανένας βέβαια να ρωτήσει αν όλα αυτά είναι αποτελεσματικά. Το θέμα είναι όμως είναι να συνεχίσουμε να αποστείλουμε αυτό το πολιτικό μήνυμα σε όλες αυτές τις χώρες χωρίς διπλά πρότυπα και χωρίς να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να καταπολεμεί την αθαντική ποινή. Ευχαριστώ κύριε Τίλεμα και σας ευχαριστώ που μας εξηγήσατε το τι γίνεται αυτή τη στιγμή μέσα στα πλαίσια του ψηφίσματος για το Ενωμένο Εθνική Συνέλευση των Εθνών. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Αρνό, εξ ονόματο τη Εκτελεστική Επιτροπή, να μα κάνει τη δική τη παρουσίαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω τονίσατε κι εσεί, εξυπακούεται ότι συνιστά αυτό προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα θεσμικά όργανά τη. Οι αρχαιότερε κατευθυντήριε γραμμέ που έχουμε είναι, δηλαδή, οι κατευθύνσει που μα δίνουν τα κράτη-μέλη για την πολιτική που ακολουθούμε για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εγκρίθηκαν το 1998 συγκεκριμένα για την θανατική ποινή. Η κυρία Άστον ε, ανέδειξε σε προσωπική προτεραιότητα αυτό το θέμα και το δήλωσε φέτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά αυτό το γνωρίζετε ήδη. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, θα ήθελα ε, να τοποθετήσω αυτό το θέμα στα πλαίσια του EAS. Ε, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συνοχή για τα μέσα που χρησιμοποιούμε και για τους θεσμικούς φορείς. Για τα μέσα, ο Μισελ Τίλεμανς μόλις μας εξήγησε τις πιέσεις που ασκούμε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τα διαβήματα για να υποστηρίξουμε αυτό το ψήφισμα που εισηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα είναι και το τρίτο του είδους. Ανέφερε επίση τα διμερεί μας διαβήματα. Πέρσι 30 το αριθμό δηλαδή ένα την εβδομάδα, ανά εβδομάδα εργασίας, κυρίως για το Ιράν και για τη ΣΥΠΑ. Θα επανέλθω μεταγενέστερα ε, για να εξηγήσω παραδείγματο χάρη γιατί έχουμε ένα τέτοιο χαοτικό κενό στην περίπτωση τη Κίνα. Επίση, ενθαρρύνουμε διοργάνωση σεμιναρίων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κρίνουμε, όπω είπε και ο κύριο Τίλεμαν, ε, να υπάρξει ευαισθητοποίηση τη κοινή γνώμη. Και αν θέλετε ε, να μιλήσετε για του πληθυσμού και για τα εθνικά κοινοβούλια, δυστυχώ πολλοί θα υποστήριζαν τη θανατική ποινή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε πανεπιστημιακό, ακαδημαϊκό επίπεδο, με, ε, από όλους τους πιθανούς διάβλους, πρέπει να εξηγήσουμε ότι αυτό το ευρωπαϊκό μέσο αυτό το μέσο, η θανατική ποινή, είναι εντελώ αναποτελεσματική, ε, πέρα από το ότι είναι παράνομη. Ε, σχετικά με το, αυτά που μας είπε ο κύριος ε, Σμιθ, εκπρόσωπος του Reprieve, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την συνδρομή σας, διότι αναφερθήκατε στο Ευρωπαϊκό Μέσο ε, για την Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Υπάρχουν 16 προγράμματα που ήδη τρέχουν στα πλαίσια αυτού του Ευρωπαϊκού Μέσου και του χρόνου θα κάνουμε προσφορά πρόταση υποβολής προσφορών για να επανεκκινηθούν οι δραστηριότητες σε αυτό το τομέα. Υπάρχουν πολλοί άριθμες δραστηριότητες, ε, κυρίως μέσα από δίκτυα, ε, όπως ε, που εκπροσωπούνται από τους συναδέλφους του πάνελ σήμερα, που δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες και καλύπτουν διάφορους τομείς, ευαισθητοποίηση της κοινή γνώμης για αυτό το θέμα, παραδείγματο χάρη μεταξύ άλλων. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όπως σας το εξήγησα, επίσης νομική αρρωγή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και παρακολούθηση των όρων εκτέλεσης της θανητικής πυρηνής, διότι γνωρίζετε ότι από Θέλουμε όχι μόνο να μειώσουμε τον αριθμό των εκτελέσεων, αλλά όταν γίνονται οι εκτελέσει θέλουμε να μεριμνήσουμε ώστε οι όροι εκτέλεση να τηρούν τα ελάχιστα πρότυπα σε διεθνέ επίπεδο ε, και κάνουμε πολλέ παρεμβάσει ούτω ώστε όσε χώρε δεν έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή ε, να περιορίσουν τουλάχιστον τη χρήση τη θανατική ποινή για τα σοβαρότερα ποινικά δικήματα και αυτό σχετίζεται με την ε, χρήση των ενόμων μέσων και της δέουσας διαδικασίας που πρέπει να ε, προσφέρεται ε, νομικά εχέγγυα, δηλαδή επιδιώκουμε για να υπάρχει ίση απονομή της ε, δικαιοσύνης που να αιτιολογεί τον αγώνα μας. Επίσης μιλήσατε για τον ιδιαίτερο ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης και τις σχέσεις που έχουμε με το Συμβουλίο της Ευρώπης. Φερρυπίν φέτος στη Λευκορωσία από με το Συμβούλιο της Ευρώπης κάνουμε ερωταστικές επαιτίους για να πείσουμε αυτό, αυτή την τελευταία χώρα με ε, ε, του ΟΑΣΑ, την τελευταία ευρωπαϊκή χώρα που διατηρεί τη θανατική ποινή, να του εντυπίσουμε να αλλάξει τη στάση της. Θέλουμε λοιπόν όλοι οι εταίροι μας να είναι αποτελεσματικοί και ε, ε, χαιρόμαστε για αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί συνιστά χειρό και ομόφωνο πολιτικό μήνυμα και νομίζω ότι εξυπακούτε πως όλοι σας υποστηρίζουν και όπως ε, σωστά είπε ο Μισελ είναι σημαντικό οι βουλευτές ως αιρετοί εκπρόσωποι του λαού αλλά και ως πολύ σημαντικά σημεία επαφής με τον πληθυσμό να συνεχίσουν αυτή την εργασία ευαισθητοποίησης τη κοινή γνώμη Τώρα η κοινωνία των πολιτών είναι σημαντική όχι μόνο επειδή προσφέρει κάποια χέγγια σχετικά με την εποπτεία, την παρακολούθηση, την νομική αρρωγή. Περνάμε μέσα από την κοινωνία των πολιτών για να υλοποιήσουμε διάφορες από τις δράσεις μας, αλλά σημαντικό είναι, ε, και σημαντικός είναι ο ρόλος τους και για τα αριθμητικά δεδομένα. Και επανέρχομαι στην Κίνα, ε, που κάνει τι ε, περισσότερε εκτελέσει και βρίσκεται κοντά στο Ιράν και στη ΣΥΠΑ. Ε, συζητούμε επί μακρόν αυτά τα θέματα στο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που κάνουμε δισετησίως με την Κίνα. Το πρόβλημα είναι ολική αδιαφάνεια ως προς τα στατιστικά δεδομένα. Δεν γνωρίζουμε τι ισχύει. Επίσης αδιαφάνεια για τις ε, διαδικασίες ε, και υπάρχει μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη εσχάτως, μια αναθεώρηση από το ανώτατο λαϊκό δικαστήριο της Κίνας σχετικά με τους όρους και τις διατάξεις περί θανατικής ποινής. Θα θέλαμε να συμμετάσχουμε στη διαδικασία, αλλά δυσκολευόμαστε όλο ιδιαίτερω ε, ω προ την πρόσβαση και την ενημέρωση για τα τεκτενόμενα στην Κίνα. Όπω ε, είπαν και οι συνάδελφοι, υπάρχουν χώρε δημοκρατικέ όπω η ΕΠΑ που μας απασχολούν, αλλά δεν μπορούμε παρά να αναφερθούμε και στην Ιαπωνία, εφόσον σα μιλάω για την Ασία. Αλλά χρειαζόμαστε μια μακρόχρονη προοπτική για την καταπολέμηση τη θανατική ποινή. Αυτό είναι σημαντικό και για τι νέε δημοσιονομικέ προοπτικέ και για την πολιτική που θα ακολουθήσουμε για το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η Ιαπωνία ξανάρχισε φέτος το καλοκαίρι της εκτελέσεις ε, και παρότι κάνουν προσπάθειες για να επικρατήσει η διαφάνεια, πρώτη φορά δηλαδή προσκάλεσαν δημοσιογράφους για να επισκεφθούν την αίθουσα των εκτελέσεων. Ξέρω πόσο ανατριχιαστικό είναι αυτό, αλλά ε, ξανάρχισαν τις εκτελέσεις και αυτό είναι κακός ιονός για την συνοχή ανάμεσα στις δράσεις όλων των εταίρων. Σας μίλησα για το, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο, για την κοινωνία των πολιτών, αλλά πρέπει να αναφερθούμε και στα κράτη-μέλη. Εν προκειμένου, πρέπει να μελετήσουμε την πρόταση που μόλις μας έκανε η οργάνωση Reprieve, Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τα διπλωματικά διαβήματα που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη-μέλη και την προξενική τους παρουσία που είναι εκτεταμένη σε διάφορες χώρες για να επιτύχουμε περισσότερα. Προς το παρόν η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφής. Ο συνάδελφος από το Μεξικό το υπενθύμησε δικαίως στα πλαίσια της Αβένα. Παρεμβαίνουμε για το ε, μεμονωμένο άτομο, όποια και είναι η εθνικότητα, το χρώμα του, το φύλλο του. Ε, είναι μια οικουμενική πολιτική για να βοηθήσουμε συγκεκριμένα άτομα. Ως προς την αποτελεσματικότητα. Θα έπρεπε λοιπόν να εξετάσουμε αυτή την πτυχή και υπάρχουν και δύο νέες, ε, νέες ιδέες. Ε, νομίζω ότι υπάρχει μια συνεργασία για την προξενική προστασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη που τώρα συστήνεται μια ομάδα που ε, έχει ε, επιληφθεί του ζητήματο για την προξενική συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι μια πρώτη ιδέα. Δεύτερον, τέσσερι φορέ το χρόνο τα σημεία επαφή για τα ανθρώπινα δικαιώματα συνεδριάζουν στην Ουάσιγκτον, ανάμεσα δηλαδή στι ε, πρεσβείες ε, και τι αντιπροσωπείε στη ΣΥΠΑ. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Δεκέμβριο και θα μπορούσε ενδεχομένω να εγγραφεί το σημείο αυτό στη μερίσια διάταξη. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η ιδέα και νομίζω θα πρέπει να την προωθήσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you so much, Madame Arnaud. I think it was delightful to hear that you're actively working. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε θερμά γιατί προσπαθείτε να συμπεριλάβετε τις ε, νέες, συνθήκ, νέες διατάξεις συνθήκης Λισαβόνας για να ενισχυθούν οι διάφορε αντιπροσωπείς Ευρωπαϊκής Ένωση ανά τον κόσμο σε ό,τι αφορά τη μάχη που δίνουν υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πώς μπορούν νέες αρμοδιότητες να χρησιμοποιηθούν και για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τις ε, παρεμβάσεις των προσκεκλημένων μας και θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Τρεις έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής ενδιαφέρον, η κυρία Γκόμες, η κυρία Λόχμπίλερ και η κυρία Λάτφορτ. κυρία Γκόμες πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά τους προσκεκλημένους μας γιατί πραγματικά η συζήτηση είναι πολύ σημαντική. Πολλά αναφέρθηκαν ήδη για την προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την κατάργηση της θανατικής ποινής. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στην ανάγκη εφαρμογής αυτού του προγράμματος προκειμένου να εντοπιστούν άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο και που έχουν κάποια σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να συνεχίσουμε την εκστρατεία μας για οικουμενική κατάργηση της θανατικής ποινής, όπως είπε ο κ. Κλάιβ Στάφορντ, καλό θα ήταν με την ανάμειξή μας στη συγκεκριμένη υπόθεση μπορούμε με τις, τα γραφεία μας που έχουμε σε χώρες που εφαρμόζουν τη θανατική ποινή και να βοηθήσουμε στην καλύτερη διαπαιδαγώγηση ε, επισημένοντας τον βάναυσο χαρακτήρα και τον άδικο χαρακτήρα ε, της θανατικής ποινής. Και το λέω αυτό με βάση την προσωπική μου πείρα. Ήμουν πρέσβης της Πορτογαλίας στην Ινδονησία και εκεί έκανα εκστρατεία προκειμένου να σώσω τη ζωή εγκολέζων που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο και ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί οι άνθρωποι στους οποίους επισήμαναν τις υποθέσεις αυτές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έπιασαν τόπο τα επιχειρήματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι θα σώσουμε κάποιους που έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι με την επιχειρηματολογία μας θα συνεχίσουμε την εκστρατεία μας για την οικουμενική κατάργηση της θανατικής ποινής. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό με την διάσωση των ανθρώπινων ζώων. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε το ψήφισμα της περασμένης εβδομάδας και την έκκλησή μας για την ε, υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος. θα πρέπει να διαρωτηθούμε κατά πόσο εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να γίνουμε και πιο αποτελεσματικοί σε αυτόν τον αγώνα. Γι' αυτό ήταν και πολύ χρήσιμη η σημερινή ακρόαση. Θα δούμε πώς μπορούμε στις επαφές μας με τις χώρες, ιδιαίτερα τις χώρες που εφαρμόζουν την ε, θανατική ποινή, πώς μπορούμε να προβάλλουμε τα επιχειρήματά μας, αλλά μπορούμε να ασκήσουμε πίεση και στο Συμβούλιο και στην υπατή εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική, να κάνουν διαβήματα προς τις χώρες που είναι απρόθυμες ακόμη και για τη συζήτηση αυτών των θεμάτων, ιδιαίτερα την Κίνα. Ξέχασα να σας πω ότι σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, το παράδειγμα του Μεξικού είναι χαρακτηριστικό. Θα πρέπει να επενέσουμε λοιπόν αυτή τη χώρα και να αξιοποιήσουμε την εμπειρία που αποκόμισε το Μεξικό από την εφαρμογή του προγράμματος. Σας ευχαριστώ. Κύριε Λόχμπιλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους όσους ε, μας κάνανε τις ε, παρουσιάσεις των απόψεων και δηλώσεων τους. Ναι, πραγματικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε μια ενιαία άποψη. Θυμίσω και την συζήτηση την περισμένη εβδομάδα, όπου ορισμένοι ε, βουλευτέ εκφράστηκαν υπέρ τους ε, ε σημασίες που μπορεί να έχει θανατική ποινή. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι λίγοι, αλλά όμως ε, υπάρχουν. Στα πλαίσια τη πρώτη ψηφίσματο υπήρχε κάτι πάνω στο οποίο δεν μπορούσαμε ομόφωνα να συμφωνήσουμε, αλλά όπου υπάρχει ανάγκη συζήτηση. Η πρόκειται παραδείγματο χάρη για το ότι στα πλαίσια τη στρατηγική να περιορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να τιμωρηθούν λόγω των εγκλημάτων τους με θανατική ποινή. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό προσεκτικά και νομίζω ότι ο εκπρόσωπο του Διεθνού Συνασπισμού κατά τη θενατική ποινή αναφέρθηκε σε αυτό. Κατά πόσο δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη προωθούν αυτά τα προγράμματα καταπολέμησης ναρκωτικών που είναι βέβαια ε, σημαντικά αλλά ίσως οδηγήσουν στο ότι σε κάποιες χώρες επιβάλλεται θενατική ποινή στους εμπόρους ναρκωτικών. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συζητήσουμε στο Κοινοβούλιο, δεν είναι εκεί να το γράψουμε δηλαδή στην πρόταση ψηφίσματο. Και τώρα που ερχόμουν εδώ υπάρχει μία μελέτη της Διεθνής Οργάνωσης Μείωσης ε, των ε, Προβλημάτων αυτών και εμείς θα μπορούσαμε να προετοιμάσουμε μία οδηγία για να μην συμβάλλουμε αυτά τα προβλήματα καταστολής του εμπορίου ναρκωτικών να οδηγούν σε θανατικές ποινές των εμπόρων. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο ε, Ραφέλ Σενουίλ Χαζάν πώς το βλέπει τα πράγματα και επίσης μια προς την Κομισιόν πόσες χώρες είναι εκείνες στις οποίες υπάρχουν αυτά τα προβλήματα της, ε, ε, κατά των ναρκωτικών και κατά πόσες χώρες αυτές επιβάλλεται θανατική ποινή ή όχι. Ευχαριστώ κύριε Λοχπίλερ, λέει η πρόεδρος. Θα ήθελα να επιβάλλω, να επιστήσω την προσοχή σε ένα σημαντικό κείμενο που έχουμε στα χέρια μας όσον αφορά την ε, ε διεθνή οργάνωση μείωσης των προβλημάτων. Και όπου Υπάρχει εκεί η αναφορά σε αυτό το ενδεχόμενο διπλό, τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που χρησιμοποιούμε. Και όπου όλο αυτό το θέμα των ναρκωτικών είναι ένα θέμα που οπωσδήποτε κάποια στιγμή που επιτροπούμε θα πρέπει να το εξετάσει σοβαρά. Τέλο πάντων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στην Σάρα Λάτφορ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την διοργάνωση αυτής της δημόσιας ακρόασης και να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ομιλητές και ιδιαίτερα τον Κλάιβ Στάφορτ Σμιθ για το πολύ ενδιαφέρον του σχέδιο γιατί ο Κλάιβ σήμερα μίλησε ως Αμερικανός αλλά έχει γραφείο της οργάνωσης του Reprieve ακόμη και στη δική μου εκλογική περιφέρεια το Λονδίνο και πραγματικά θα ήθελα να τον επενέσω για την καταπληκτική δουλειά που κάνει η οργάνωσή του, ρίπριβαλε και ο ίδιος. Επίσης, ε, ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο από το Μεξικανικό Προξενείο. Αλλά ε, βέβαια το Μεξικό δεν είναι χιλή, αλλά όλα τα ισπανικά που ακούσαμε το τελευταίο 24 ώρα από τη χιλή και πώς α, ε, πριτάνευσε η η αγάπη για την ανθρώπινη ζωή, για, χάρη στη διάσωση των αποκλωβισμών των 33 μεταλλορίχων, γιατί μίλησε για σχιζοφρένεια ο Κλάιβ, αλλά πραγματικά μείναμε προσκολλημένοι στις οθόνες της τηλεόρασης περιμένοντας τη διάσωση αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, έχουμε εδώ δύο διαφορετικά πράγματα. Έχουμε την πολιτική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ιδιαίτερα δραστήρια και μάλιστα και επιτυχής σε ό,τι αφορά τις πιέσεις που ασκεί. Βέβαια, η αξιοπιστία που έχουμε επιτυχεί δεν είναι πλήρης ακόμη και διαπιστώνω ότι η Λετωνία δεν έχει ακόμη καταργήσει πλήρως την θανατική ποινή. Ελπίζω να μην κολλήσει η ε, για κάτι τέτοιο και εγώ ελπίζω ότι όλες οι χώρες που προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταργούν προηγουμένως ε, τη θανατική ποινή. Αλλά φαίνεται ότι η Λετωνία την ε, διατηρεί για ορισμένα πολύ σοβαρά εγκλήματα. Ήταν πολύ συγκεκριμένα και πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε ο Κλάιβ, αλλά και τα καταληκτικά σχόλια της κυρίας ε, Άρνο. Και με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ελπίζουμε ότι θα βελτιωθεί ο συντονισμός και θα έχουμε πιο κοινέ δράσεις των ευρωπαϊκών χωρών, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συντονιστεί και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τώρα που ως ε, συμβαλόμενο μέρος θα προσυπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με δική της νομική προσωπικότητα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την ύπατη εκπρόσωπος ε, One Stop Shop ως ε, σημείο επαφής ε, για τις επαφές με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που θα ειδοποιούν την, το γραφείο της ΥΠΑ της εκπροσώπου για πιθανές απειλέ ή καταδίκες σε θανατική ποινή, ώστε να λαμβάνονται κεντρικά αυτές οι πληροφορίε από το γραφείο της ΥΠΑ της εκπροσώπου Βρυξέλλες και να μπορούν συνέχεια να διαβιβάζονται στις ενδιαφερόμενες κυβερνήσει, ώστε να είναι πολύ πιο συντονισμένη και η απάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με συγκλώνηση και ομολογώ εδώ την ε, άγνοιά μου η παράθεση ε, της ε, δήλωσης ε, της, του Ευρωπαϊκού Υπουργείου Εξωτερικών σε ό,τι αφορά τα προξενικά καθήκοντα και τη δυνατότητα εκπροσώπησης των αλλοδαπών υπηκών. Πραγματικά δεν παρακολούθησα ούτε τις εξελίξεις στην EEAS, του ε, τους ε, κανονισμούς, δηλαδή λειτουργίες για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράσης και ποια πραγματικά θα είναι τα καθήκοντα της ε, εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τέτοιες περιπτώσεις. Από ό,τι ξέρω και η Χίλαρη Κλίντον είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Μπούζα και τη συνδιάσκεψη των πρόεδρων. δυστυχώς ε, παρόλο που είμαι αντιπρόεδρος, πρώτη αντιπρόεδρος στην ε, κοινοβουλευτική αντιπροσωπή για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, δεν με εξασφάλισε πρόσκληση για συνάντηση με την κυρία Χίλαρη Κλίντον. Δεν, θα δεν μπορώ, μπορώ καν να παραστώ στις συναντήσεις που θα έχει με τη διάσκεψη των Προέδρων. Πάντως θα μπορούσαμε να έχουμε μια ένα καλύτερο συντονισμό και καλύτερη διασύνδεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, με ιδιαίτερη επικέντρωση σε αυτά τα θέματα. Έχουμε δικαστική αρρωγή στα θέματα έκδοσης, έχουμε προγράμματα για διαβίβαση δεδομένων ή κοινή χρήση δεδομένων. Γιατί λοιπόν ε, να μην έχουμε και μια κοινωτική στρατηγική για την παροχή αρρωγής σε Ευρωπαίου υπηκόου που έχουν εμπλακεί στα γρανάζια του δικαστικού συστήματο των Ηνωμένων Πολιτειών ή άλλων χωρών. Γιατί όλα πάνε καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι ότου βρεθούμε μπροστά στην πρόκληση του συντονισμού. Υπάρχουν και διεθνείς συμφωνίες, ε, διεθνείς συμφωνίες συνεργασίες ε, ή συμφωνίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί να μην ενημερωνόμαστε καλύτερα όταν συλλαμβάνεται ένας Ευρωπαίος επίκος ή ε, κατηγορείται σε μία από τις χώρες αυτές. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που είναι άγνωστες για το πώς λειτουργούν αυτές οι συμφωνίες που έχουμε με τρίτες χώρες. Επίσης, η μελέτη της ε, οργάνωσης Reprieve είναι πολύ χρήσιμη να χαράξουμε μια πανευρωπαϊκή στρατηγική που θα αντικαταστήσει αυτές τις ε, μεμονωμένες προσεγγίσεις που γίνεται, που είναι πολύ εγκατασπαρμένες. Έχουμε μια ενιαία υπηρεσία εξωτερικής δράσης, έχουμε ψήφισμα. Γιατί λοιπόν να μην έχουμε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έναν ενιαίο οργανισμό αντίδρασης, απόκριση της περιπτώσεις. Ευχαριστούμε, Εμιλή. Είπατε ότι πρόκειται για ένα εργαστήριο. Ναι, τελικά εργαστήριο έχουμε γίνει για να ανακαλύψουμε πώ μπορούμε να ενισχύσουμε την εκστρατεία για την ε, κατάργηση της ε, θανατική ποινή. Χαίρομαι που παρίστανται πολύ σημαντικοί φορείς και από την κοινωνία των πολιτών και από τα θεσμικά όργανα και από το διπλωματικό σώμα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σα Είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο κύριος Τίλεμας και η κυρία Αρνό σίγουρα θα θέλουν να δευτερολογήσουν μετά από όλε αυτέ τις ε, που ακούστηκαν ε, επί τη βάση των ε, εισηγήσεων του κυρίου Στάνφορντ. Η κυρία Ντεκέιζερ τώρα. Ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη γιατί πολλά τα είπαν ήδη οι συνάδελφοι και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Κυρίως για τις ε, διάφορες παρεμβάσεις ε, που ακούσαμε νωρίτερα. Μιλήσαμε για το θέμα της ευαισθητοποίησης ε, της κοινή γνώμης ε, για τη θανατική ποινή. Αναρωτηθήκαμε τι να κάνουμε, πώς να δράσουμε σε επίπεδο κυβερνήσεων, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών για να βοηθήσουμε τους επικούς των χωρών μας. Αλλά δεν μιλήσαμε καθόλου για τη σύναψη των συμφωνιών από πλευρά τη Ένωση και πώς μπορούμε μέσα από αυτή την εξουσία που έχουμε στα χέρια μας ε, με αυτές τις συμφωνίες, τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε τον αγώνα κατά της θανατικής ποινή και να προωθήσουμε το θέμα του μορατόριου. Υπάρχει η παράγραφος 15 στο ψήφισμα που ζητείται από, το Κοινοβούλιο και το, ε, από την Επιτροπή και το Συμβούλιο όταν συνάπτουμε μία συμφωνία να θέτουν το ζήτημα τη κατάργηση τη θενατική ποινή και να ενθαρρύνουν τα κράτη-μέλη με τα οποία συνάπτουν συμφωνίε, αν δεν το έχουν ήδη κάνει, να καταργήσουν ή να περιορίσουν τη χρήση τη θανατική ποινή. Ε, γίνονται αυτές οι προσπάθειε ποιε είναι οι επιτυχίε που έχουν σημειωθεί, ε, ε, μιλάμε σήμερα για τη χρήση αυτών των μέσων που έχουμε, τις εμπορικές συμφωνίες, συμφωνίες εταιρικής σχέσης, ούτως ώστε να σημειωθεί πρόοδος ε, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Τι γίνεται όμως με τη θανατική ποινή, τι έγινε, τι έχουμε καταφέρει. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Και δεύτερον, χώρες όπως η Ιαπωνία και άλλες επανέρχονται, ε, επανισάγουν την ε, θανατική ποινή ε, έχοντας ένα όσο είδους ε, opting out για την τρομοκρατία ε, ή για τα ναρκωτικά, χρησιμοποιώντας δηλαδή τη θανατική ποινή σε αυτές τις περιπτώσεις. Μα είναι αν, ανησυχητικό γιατί αυτό αντιβαίνει στις σημερινές τάσεις και μην ξεχνάμε ότι με την σημερινές συγκυρίες θα μπορούσε να υπάρξει εκτεταμένη επανεισαγωγή του θεσμού της θανατικής ποινή, σε ειδικέ όπως χαρακτηρίζεται περίπτωση. Ευχαριστούμε κύριε Ντεκάισε αυτό το θέμα των Διεθνών Συμφωνιών Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτε χώρε είναι μεγάλη βαρύτητα για το Κοινοβούλιο και για την υποεπιτροπή μα συγκεκριμένα, κυρίω τώρα που το Κοινοβούλιο έχει νέε αρμοδιότητε μετά τι συνθήκε Λισαβόνα, μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει διεθνεί συμφωνίε. Και το θέμα τη ρήτρα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξετάζεται διεξοδικά ε, σήμερα και ε, σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες που έχουμε για την κατάργηση θανατικής Ποινή. Ο κύριος Κροζέτα έχει, είναι ο τελευταίος ομιλητής. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρωτοβουλία κατά τη γνώμη μου, διότι ε, οφείλουμε να εξετάσουμε αυτό το θέμα. Ε, το, κυρίως τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη θανατική ποινή και το ε, θέμα των ναρκωτικών. Δηλαδή η χρήση της θανατικής ποινής για αδικήματα που ε, σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Σε τι έγκυται αυτό κυρίως στην κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Κάποιες χώρες εφαρμόζουν την θανατική ποινή για κατοχή μικρής ποσότητας ακόμη και κάναβης ή άλλων ναρκωτικών ουσιών Ήμουν στην ε, Σαουδική Αραβία στην πρώτη αποστολή που έκανα και στο αεροπλάνο μου έδωσαν ένα έντυπο να συμπληρώσω όπου έλεγε πως ε, ε, οφείλω να δηλώσω ότι δεν έχω στην κατοχή μου ε, ναρκωτικές ουσίες και να αναγνωρίσω ότι η απλή κατοχή ναρκωτικών ουσιών ε, τιμωρείται με τη θανατική ποινή στη Σαουδική Αραβία και δεν είναι η μόνη χώρα στον κόσμο η Σαουδική Αραβία που χρησιμοποιεί ε, τις καταδίκες αυτές στο αεροπλάνο λοιπόν σκέφτηκα αυτοί οι νέοι που ε, ταξιδεύουν ε, προς και διέρχονται από τη Σαουδική Αραβία. Ε, ορισμένοι λοιπόν ε, συλλαμβάνονται ή και θανατώνονται. Πρέπει να υπερασπιστούμε λοιπόν την ανθρώπινη ζωή. Οι έμποροι ναρκωτικών φέρνουν το θάνατο και τιμωρούνται. Δηλαδή χρησιμοποιείται αυτό ως μέσο καταστολής, ε, βάναυσης ε, συμπεριφοράς ε, και θανάτου, επιβολής θανάτου. Ε, Ε, εγώ δεν θέλησα να συνεχίσω να συνεργάζομαι με τη Σαουδική Αραβία που τόσο κατάφορο παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, σε μία εκπομπή στην τηλεόραση παρακολούθησα ε, μία εκτέλεση γιατί ε, σε αυτή τη χώρα υποχρεούνται ε, οι πολίτες ε, να παρευρίσκονται στις εκτελέσεις, εφόσον βρίσκονται στο χώρο της εκτέλεσης, Ε, και στη ΣΥΠΑ η διαδικασία εκτέλεσης παίρνει μόνο λίγα δευτερόλεπτα, αλλά αυτό δεν σημαίνει Σαουδική Αραβία. Χρησιμοποιούν μαχαίρες ε, που, ε, και καταφέρνουν χτυπήματα, πολλαπλά χτυπήματα στο σβέρκο των θυμάτων και ο Δήμιος επαναλαμβάνει αυτά τα χτυπήματα ε, είναι μια πρακτική τρέχουσα σε πολλές χώρες της Εγγύης και Μέσα Ανατολής. Ε, είναι απίστευτο, δημιουργεί εκδικητικές ε, τάσεις. από τις Φιλιππίνες υπήρχε ένας ομοφιλόφιλος Νέλ Τουρμπό που εκτελέστηκε το 1995 και υπήρχε και δικαστικό λάθος δεν ξέρω αν γνωρίζετε την υπόθεση. Είχε βρεθεί νεκρή μία γυναίκα που συνεργαζόταν με αυτόν τον νέο Φιλιππίνο ομοφιλόφιλο και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες χρησιμοποίησε ως μάρτυρα τον φίλο του ε, γιατί όταν ε, δολοφονήθηκε η γυναίκα βρισκόταν με το φίλο του ε, μετά από ένα χρόνο σε μία φυλακή με βαδό ένα επί 1,5 μέτρο Περίμενε... Το πρότυπο μας σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να είναι πολύ διαφορετικό ε, η Ευρώπη εκπροσώπησε πολύ, ε, με, με, πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα αυτά, αυτή τη θέση. Δεν επιτρέπεται να επιβάλλεται η θανατική ποινή είτε για ε, τρομοκρατία είτε για εμπόριο ναρκωτικών ε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε εδώ εφαρμόζεται και δεν εφαρμόζεται, προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε μετά για άλλα εγκλήματα βία γιατί έτσι μπορεί ίσως κάποιος να ε, προσπαθήσει να επιβάλλει τη θανατική ποινή κατά των ε, πολιτικών του παραδείγματος χάρη αντιπάλων, να κατηγορήσω εγώ τον αντίπαλό μου ότι κάνει εμπόριο ναρκωτικών ή τι, μπορεί να φροντίσω να εκτελεστεί. Ε, δεν επιτρέπεται λοιπόν να υπάρχει αυτή τη δυνατότητα. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αποφασισμένοι, θα πρέπει πραγματικά να είμαστε πάρα πολύ απόλυτοι για αυτό που κάνουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες επιβάλλουν τη θανατική ποινή, παραδείγματος χάνουν χώρες ε, παραγωγή πετρελαίου και δεν τις κατηγορούμε καθόλου αυτές τις χώρες. Ε, γιατί για με τις αραβικές χώρες υπάρχουν ορισμένες που είναι πιο μετροπαθείς, ίσως και μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί τους, αλλά και εκεί υπάρχουν ακραίοι ε, προασπιστές ε, της θανατικής ποινής. Και πολλές φορές αυτές οι καταδίκες είναι, χώρες, είναι πρόσωποι από χώρες όπως την Ινδία, το Πακιστάν κλπ. που είναι στις ε, χώρες τις ε, αραβικές είναι σκλάβοι είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται εκεί, τους παίρνουν το διαβατήριο, δεν μπορούν να φύγουν, δεν μπορούν να αντιδράσουν, είναι σε μια κατάσταση πραγματικά σκλαβιάς εκεί. Όλα αυτά είναι θέματα που θα πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινίσουμε και για την περιοχή αυτή. Ακόμα και το θέμα του ορισμού και το θέμα της, του πολι... της παράδοσης αυτής της βίας που δεν υπάρχει μόνο στο Ιράν. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Οπωσδήποτε χρειάζεται να αποδώσουμε μεγαλύτερη σημασία στις χώρες ε, του Περσικού κόλπου και της Μέσης Ανατολής. Γιατί υπάρχουν σημαντικές παρέμβασεις ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η θανατική ποινή. Εδώ κλείνω τον κατάλογο των ε, συναδέλφων που θέλουν να μιλήσουν. Ξαναρχίζω όμως με τους επισκέπτες μας. Αρχίζω με τον κύριο Σταφάρτ Σμιθ ισως δυο δύο-τρία λεπτά να μπορείτε να αρκεστείτε γιατί έχουμε βέβαια τη δυνατότητα να σας δώσουμε το λόγο και στις μία στην ε, συνέντευξη τύπου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνικός. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα σχόλια που ακούσαμε. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων χωρών, όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι Μεξικανοί μας βοηθούν και με Βρετανούς υπηκόους που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο στο Τέξας. Οπότε υπάρχει συνεργασία, όπως μας είπε πριν και ο εκπρόσωπος από το Μεξικό. Σάρα, το ίδιο συνέβη με τους, ε, με τους Οι Μεξικανοί με παρόμοιο τρόπο ε, σώζουν ζωέ ανθρώπων που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο στις Ηνωμένε Πολιτείε. Αλλά και για τα ναρκωτικά. Θα ήθελα να πω ότι στο Λαός εκπροσωπήσαμε μια γυναίκα που είχε καταδικαστεί και το λαό επικαλέστηκε την ε, συνθήκη για την καταπολέμηση των ναρκωτικών που λέει οφείλετε να τιμωρήσετε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, ότι οφείλετε να τιμωρήσετε, δεν σημαίνει ότι είστε υποχρεωμένο να εφαρμόσετε κατά δίκη θανατική. Και Πρόκειται για σύμβαση του ΟΗΕ, γι' αυτό και θα πρέπει να αποφύγουμε γελίες ερμηνείες συμβάσεων του ΟΗΕ, γιατί πολλές φορές επικαλούνται διατυπώσεις για να τεκμηριώσουν τη θέση τους. Και είμαι σαφώς υπέρ του One Stop Shop στις Βρυξέλλες, να υπάρχει ένα ενιαίο γραφείο που θα συγκεντρώνει τις πληροφορίες. Και σε συνεργασία με τους συναδέλφους και του Παγκόσμιου Συνασπισμού κατά της θανατικής ποινής, καλό θα ήταν να συντονιστούμε και μακάρι να έχουμε εδώ ένα ενιαίο γραφείο ώστε να μπορούμε να έχουμε τη συνεργασία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ενημερώνεται για τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα το θέμα της ε, νομοποιημένης επέμβασης ευρωπαϊκών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ασχοληθούμε την επόμενη εβδομάδα αυτό το θέμα των ε, εκτελέσεων high-tech στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ε, υπάρχουν ε, συγκεκριμένες εταιρείες που παρασκευάζουν τα ναρκωτικά που χρησιμοποιούνται στις θανατικές εκτελέσεις. Και ίσως θα υπάρχουν σχετικές διατάξεις που θα απαγορεύουν σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε, τέτοιους, σε τέτοιες διαδικασίες. Πάντως είναι πραγματικά πολύ ελκυστική αυτή η προσπάθεια περαιτέρω συνεργασίας για την εφαρμογή όλων αυτών των πρωτοβουλειών για την καταπολέμηση της ε, θανατικής ποινής. Ίσως τέτοιου είδους ναρκωτικό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ε, εργαλείο βασανισμού γιατί έχουμε σχετική νομοθεσία εις βάρος ε, κατασκευαστών τέτοιων εργαλείων βασανισμού. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος ε, Ραφαέλ Σενέχασαν. Θα μιλήσω γαλλικά αυτή τη φορά. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα των ναρκωτικών και των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται μάλλον για την ε, εκτέλεση. Πολλές χώρε στην Ασία, αλλά και στον αραβικό κόσμο, καταδικάζουν και εκτελούν ανθρώπους μόνο και μόνο για απλή κατοχή ναρκωτικών ή για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, όπω μα είπε κάποιος ευρωβουλευτής ε, για την κατοχή στην Σαουδική Αραβία μπορεί να τιμωρηθεί κάποιος για θανατική ποινιά και σε άλλες ε, αραβικές χώρες. Πραγματικά είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια και πολλές από τις χώρες αυτές είναι και τουριστικοί προορισμοί. Είναι χώρες με τις οποίες έχουμε στενές εμπορικές σχέσεις και εμπορικές συμφωνίες με τέτοιες αραβικές χώρες. Θα μπορούσαμε λοιπόν ε, να εξετάσουμε περαιτέρω αυτή την κατάσταση και να υιοθετήσουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Και η δεύτερη τάση που ανέφερα και προηγουμένως είναι αυτή η προσπάθεια εύλογου αγώνα και καταπολέμησης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έχουμε και μια σχετική μελέτη που ήταν πολύ χρήσιμη αλλά ταυτόχρονα Ορισμένες χώρε που δεν εφαρμόζουν σήμερα τη θανατική ποινή δεν τη χρησιμοποιούν πια έχουν τάση να την επαναφέρουν ε, προκειμένου να καταστήσουν πιο αποτελεσματικό τον αγώνα τους ε, κατά των ναρκωτικών. Και αυτό δεν το παρατηρούμε μόνο στην Ασία και τον Αραβικό κόσμο. Δυστυχώς ε, το βλέπουμε και στη Λατινική Αμερική, Κεντρική και Νότια Αμερική. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τίλεμος, τώρα και κατόπιν η κυρία Αγνώ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω κι εγώ αποκλειστικά γαλλικά. Μα ναι, πολύ καλά κάνετε. Βεβαίω, γιατί είναι και σαφέστερο και έχετε και τέλειου διερμηνεί. Ευχαριστούμε εκ μέρου του μιλητή. Πρώτο σημείο, αυτό το σχέδιο, αυτό το πρόγραμμα που ε, ενδέχεται να προταθεί για την ε, προξενική συνεργασία των κρατών μελών. Ε, λίγα είναι ενδιαφέρον το θέμα και η κυρία Αχνό σίγουρα θα έχει πολλά στοιχεία να προσθέσει, διότι εισερχόμεθα προκειμένου σε ένα τομέα όπου υπήρχε μικρότερο συντονισμό σε σχέση με άλλους τομείς της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε ενδεχομένω ε, να εξετάσουμε σε μεταγενέστερο στάδιο και υπό το φως της συνθήκης της Λισαβόνας ε, τα όσα είναι εφικτά σήμερα πλέον. Γιατί όπως γνωρίζετε στο παρελθόν αυτές οι πολιτικές, και το, έχω, και το είπα ήδη, ε, δεν έτυχαν μεγάλου συντονισμού. Υπάρχουν και κάποιες ευαισθησίες από πλευράς κάποιων μελών και πρέπει να τις λάβουμε υπόψη και να συνε... Ε, με προξενικά μέσα κάποιες κυβερνήσεις θέλουν να προστατεύσουν τους υπηκόους τους. Υπάρχει μια δυναμική και πρέπει να την ενισχύσουμε. Πάντως ε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι υπάρχει μια αδύρυτη ανάγκη να ενισχύσουμε και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό, πέρα από αυτά που κάνουν τα κράτη-μέλη. Για την καθυστέρηση που σημειώνεται η κυρία Ντικέιζερ μας μίλησε για την Ιαπωνία συγκεκριμένα. Λοιπόν, μία λύση είναι να υπερασπιστούμε την επικύρωση του δευτέρου προαιρετικού πρωτοκόλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Τι προβλέπει το πρωτόκολλο κατάργηση της θανατικής ποινής. Ιδού λοιπόν ένα μέσο του ΟΗΕ. Ε, επί του οποίου με πυγμή μπορούμε να βασιστούμε ε, και να ε, βασίσουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Πολλά κράτη-μέλη, γνωρίζετε, έχουν ήδη υπερασπιστεί ένθερμα την επικύρωση του πρωτοκόλλου αυτού, μεταξύ των οποίων και το Βέλγιο. Και για να σας μιλήσω και λίγο για τη χώρα μας, ένα πενευτό, ένας Βέλγος ε, συνέταξε αυτό το δεύτερο προαιρετικό πρωτόκολλο. Τέλος φανώ με την ιδιότητα του Προέδρου της ΕΚΟΧΟΜ, τονίζω ότι από το φετινό φθινόπωρο έχουμε πλέον αυξημένη πεποίθηση σχετικά με το ότι θα προχωρήσει η Ένωση ως Ένωση για να τονώσει τις εκστρατείες υπέρ της επικύρωσης αυτού του δευτέρου πρωτοκόλλου, κυρίως την εκστρατεία της παγκόσμιας, ε, του Παγκόσμιου Συνασπισμού κατά της θανατικής ποινής που εκπροσωπείται εδώ σήμερα. Τρίτη παρατήρηση για το θέμα των ναρκωτικών ε, και τη σχέση τους με τη θανατική ποινή ένας από τους ομιλητές ε, χρησιμοποίησε το επίθετο γελίος. Μα είναι πολύ εύστοχο. Είναι γελίο, όντως. Ε, σε αυτό το τομέα ερμηνεύονται έτσι οι διατάξεις ώστε να επιτρέπεται η θανατική ποινή. Μα αυτό αντιβαίνει στο ίδιο το ένομο μέσο που χρησιμοποιούν ε, στον ΟΗΕ, δηλαδή, με, χάρη σε αυτό το δεύτερο προαιρετικό πρωτόκολλο. Ε, ε, προφανώς είναι εσφαλμένη η ερμηνεία στα μάτια του Γενικού Γραμματέα του και της Γενικής Συνέλευσης του ΙΔΟΥ. Ευχαριστούμε κύριε Τίλε ε, και συγχαρητήρια προς το Βέλγιο γιατί συντάξατε το δεύτερο προεδρικό πρωτόκολλο. Κυρία Άγνο, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να απαντήσω στην κυρία Ντεκάιζερ. Δηλαδή, ε, στις συμφωνίες που συνάπτουμε με τρίτες χώρες, αν μπορούμε να έχουμε ε, μια προϋπόθεση, για τη, μια ρήτρα δηλαδή για τη θανατική ποινή. Όχι, ποινή. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί δεν είναι παράνομο πλευρά διεθνού δικαίου. Επιτρέπεται για τα σοβαρά ποινικά δικήματα. Εκτό, όπω εξήγησε και ο Μισελ, αν κάποια χώρα έχει επικυρώσει το δεύτερο προαιρετικό πρωτόκολλο πιστεύουμε Εφόσον υπάρχει ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στι περισσότερε συμφωνίε και μέσω αυτού ε, ε κατοχυρώνεται ένα διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουμε ένα σημείο εισόδου και μπορούμε έτσι να πιέσουμε για την κατάργηση τη θανατική ποινή ή τουλάχιστον ε, να ενθαρρύνουμε τον περιορισμό στη χρήση τη θανατική ποινή. Και όταν μα ρωτάτε αν θεωρούμε πω έχει σημειωθεί πρόοδο με τέτοιου είδου πιέσει, κοιτάξτε, από πλευρά διαλόγου το Τογκό και οι Φιλιππίνε είναι χώρε όπου μπορέσαμε να δράσουμε αποτελεσματικά. Για τα ναρκωτικά, όπως ακούσαμε ήδη, είναι σαφές ε, πως ε, οι εκτελέσεις που συνδέονται με τα ναρκωτικά, μάλλον να το πω αλλιώς, δεν θεωρούνται τα ναρκωτικά ως ε, ποινικό αδίκημα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό ως νομικό επιχείρημα, αλλά μας ανησυχεί, όπως είπε και ο κύριος Κορτσέτα, ε, ότι κάποιες χώρες ε, χρησιμοποιούν τη θανατική ποινή για ε, αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Είμαστε σε επαφή με διάφορες χώρες, ειδικά για αυτό Ινδονησία, Ταϊλάνδη, Γκάμπια και όπως είπε και η κυρία Γκόμες και η κυρία Λάτφορντ σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε για το θέμα των ναρκωτικών, ένα πράγμα που μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό είναι το εξής. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης που προσαρμόστηκε πέρσι το Δεκέμβριο το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο τομέα της ελευθερίας δικαιοσύνης και της ασφάλειας. Έτσι. Σε αυτό το πρόγραμμα της Στοκχόλμης υπάρχει δέσμευση ε, βάσει της οποίας ε, πρέπει να εξεταστεί ο αντίκτυπος Τη εξωτερική δράση τομέα δικαιοσύνης ε, ε, και της ασφάλειας, ε, λαμβάνοντας υπόψη την πτυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εκεί συμπεριλαμβάνεται και η θανατική ποινή. Δηλαδή, όταν εφαρμόζεται εξωτερικά αυτή η δράση, πρέπει να εξετάζουμε ποιο είναι ο αντίκτυπο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό τι σημαίνει ότι σε κάποιο στάδιο μπορούμε να εξετάσουμε και την συνδρομή στα διάφορα προγράμματα καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών, ναρκωτικών. Δηλαδή υπάρχει μια πολιτική πτυχή που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Κάτι άλλο. Έχουμε εδώ τον επικεφαλής του προγράμματος. Λοιπόν, ε, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που μόλις τώρα άρχισε Ε, από την οργάνωση, διεθνή οργάνωση μείωσης ε, των ζημιών ε, όπου εξετάζεται αυτή ακριβώς η πτυχή, δηλαδή η σχέση της επιβολής θανατικής ποινής με τις διεθνείς προσπάθειες καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών και επιβολής των σχετικών νομοθεσιών. Τρίτον, χαίρομαι πάρα πολύ που μου καλέσατε σήμερα, γιατί αύριο θα γίνει ετήσια διαβούλευση στη Βιέννη ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ και θα μπορέσω εγώ αύριο στη Βιέννη να το αναφέρω αυτό όταν ασχοληθούμε με το θέμα των ναρκωτικών και επίσης υπάρχει ένα ευρύτατο πρόγραμμα συνεργασίας με την ε, ε, UNDC, την ε, υπηρεσία του ΟΗΕ. Μάλιστα λέει η Πρόεδρο. Σας ευχαριστούμε. Ε, ε, αναφερθήκατε στον εκπρόσωπο της Διεθνούς Οργάνωσης Harm Reduction. Βρίσκεται εδώ στην αίθουσα και προσπάθησαν ε, να καλύψουν διάφορα προβλήματα που προανέφεραν οι συνάδελφοι. Οπότε θα μπορούσε ο εκπρόσωπο αυτής τη οργάνωσης να πάρει το λόγο και να μας μιλήσει για λίγα λεπτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το εκτιμούμε. Τώρα αρχίζουμε τη συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα απορίσματα της μελέτης που κάνουμε. Ε, παρουσιάσαμε τις ε, συστάσεις μας ε, και έτυχαν θετικής αποδοχής και συνεχίζονται οι συζητήσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα που εντοπίσαμε. Πολλά προγράμματα κατά πολέμηση των εμπορίων ναρκωτικών θεωρούνται ως αυτός σκοπός. Όσα κιλά και αν κατάσχουμε, όσοι και αν συλληφθούν δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όμως υπάρχει μια σκιά, η θανατική ποινή ε, και είναι ανησυχητικό αυτό σε σχέση με την επιτυχία μπορεί να σημειώσει κάθε τέτοιο πρόγραμμα. Δηλαδή, προγράμματα που εφαρμόζουν, ε, εφαρμόζονται από την αρμόδια υπηρεσία ε, του ΟΗΕ μπορούν να λαμβάνουν υπόψη αυτή την πτυχή της θανατικής ποινής, ε, ούτως ώστε εξ αρχής σε προγράμματα επιβολής νόμου και καταπολέμησης των εμπορίου ναρκωτικών να λαμβάνεται υπόψη αυτή η πτυχή σε επίπεδο προγραμματισμού ή και υλοποίηση. Επίσης, πώς οι δωρητές όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να συμβάλλουν λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε εξ είτε παρέχοντας συγγνώμη, υποστήριξη ε, ε, όσο τρέχουν τα διάφορα προγράμματα. Και συνεχίζονται και τα προγράμματα και οι συζήτησεις. Αυτά. Σας ευχαριστούμε για την ε, επί τούτο παρουσίαση της οργάνωσής σας ε, και τις σχέσεις που έχετε με την ε, καταπολέμηση θανατικής ποινής. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Όντως, σήμερα κάναμε ένα εργαστήριο για τις κοινέ προσπάθειες για την της θανατικής ποινής. Ελπίζω ότι αυτό θα οδηγήσει σε αυτά αποτελέσματα Φυσικά θα λάβουμε υπόψη όλες τις προσπάθειες και τις προτάσεις που διατυπώθηκαν από τους επιφανείς προσκεκλημένους μας και τις προτάσεις με κυβερνητικών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών αλλά και των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Θα ήθελα εδώ να ολοκληρώσουμε τη δημόσια ακρόαση. Ο κύριος Κλάιβ Στάφορντ Σμιθ, περίπλοκο το, ένα, το όνομά σας, δεν μπορώ να το θυμάμαι απ' έξω. Ο κύριος Κλάιβ Στάφορντ Σμιθ μίλησε ιδιαίτερα για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να σώσει τους καταδικαστέντες σε θάνατο Ευρωπαίους πολίτες σε διάφορες ε, χώρες του κόσμου. Και ε, νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία που προαναγγέλλεται. Τώρα η πρόταση μου μέχρι τις 12.30 είναι να συζητήσουμε με τον επιφανή μας προσκεκλημένο από το Ιράν και συζήτηση παρουσία του Προέδρου της ε, ειδικής αντιπρο... κοινοβουλευτικής αντιπροσωπής για τη σχέση με τον Ιράν προσκάλεσε και τον ε, εκπρόσωπο από το Ιράν. Επίσης έχουμε και την ε, εξέταση γνωμοδότησης για τον κανονισμό της Frontex με τεράστιες διαστάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω τον κύριο Μοχάμετ Μοσταφά Αρή που είναι ο δικηγόρος της κυρίας Σακινέα Εμάν. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συστάσεις για την κυρία Σακινέ Αμάνη, Μοχάμετ Αστιάνη. Ε, καταδικάστηκε σε θάνατο διαλυθοβολισμού μετά από ε, ποινή 99 χτυπημάτων με μαστίγιο σε δίκη που έγινε στην οποία δεν καταλάβαινε καν τη γλώσσα και δεν είχε κάνει δικαίωμα υπεράσπισης. Και μάλιστα θυμάμαι ότι μετά τη συζήτηση στην Ολομέλη της υπόθεσής της ε, καταρτήσαμε ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που σας το έχουμε μοιράσει και θα ήθελα να υπενθυμίσω τα λόγια του Πρόεδρου Μπούζεκ και τα δικά μου που επισημάναμε ότι έχουμε σοβαρές ανησυχίες για την υπόθεση αυτή και η κατάσταση όταν γνωστοποιήθηκε και καταγγέλθηκε δημοσίως ε, πήρε μεγάλες διαστάσεις. Υπάρχουν βέβαια αντικρουόμενες πληροφορίες για περαιτέρω αποφάσεις ε, περί της τιμωρίας της και πριν από δύο μέρες λάβαμε πληροφορία ότι, κυρία ο γιος της κυρία Σακινέ και ο δικηγόρος της ε, συνελήφθησαν. Ε, επανέρχομαι στον προσκεκλημένο μας τον κύριο Μοχάμετ Μοσταφάη που είναι πολύ γνωστός Ιρανός ε, συνήγορος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει υπερασπίσει δεκάδες, ε, ιδιαίτερα ανήλικους ε, κατηγορούμενους που απειλούνται με θανατική ποινή. Δυστυχώς η επιδόση του Ιράν στον τομέα αυτό είναι θλιβερές. Ο κύριος Μοχάμετ Μασταφάη θα μας κάνει μια σύντομη επισκόπηση της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν υπό το φως της νομικής κατάστασης. Καταρχήν έχουμε την σημαντική ισχύ των, των Ισλαμιστών ηγετών ε, απέναντι σε ένα πολύ αδύναμο δικαστικό σύστημα ή τη δυνατότητα των οικογενειών που έχουν προσβληθεί, που δικαιούνται ακόμη και όταν δεν προβλέπεται αυτό από τον νόμο, να ζητήσουν θανατική καταδίκη του κατηγορουμένου. Και άλλα τέτοια θέματα θα μας τα αναλύσει ο κύριος Μοχάμετ Μοσταφάη, που μας τιμά ιδιαίτερα με την παρουσία του και χαίρομαι γιατί θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις της υπόθεσης Σακινέ Μοχαμαντία Στιάνη, αλλά και και τις ε, διάφορες λεπτομέρειες για τοπικό και γενικό δικαστικό σύστημα στο Ιράν. ممنون e, Σας ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας ενημερώσω για ορισμένα από τα προβλήματα ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα που διαπιστώνονται στο Ιράν και να σας δώσω και περισσότερες πληροφορίες για το πώς αντιμετωπίζει το Ιράν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα παγκοσμίω είναι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό σε όλες τις χώρες. Η τρίτη χιλιετία θα είναι η χιλιετία που θα προσπαθήσει να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν θα επικυρώνει, θα, θα θελοτυφλεί μπροστά σε καταστρατηγήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βέβαια έχουμε και συναφή προβλήματα έλλειψη ελευθερίας, έλλειψη ασφάλειας που οδηγούν σε δικτατορία, σε φονταμεταλισμό, σε τρομοκρατία και δυστυχώς οι ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι από τους πιο κατάφορους παραβιαστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων εγκρίνουν λιθοβολισμού σε θάνατο, γίνονται αυθαίρετες εκτελέσεις, ακόμη και μαζικές εκτελέσεις, πολιτικές εκτελέσεις, εκτελέσεις ανηλίκων, ατόμων κάτω των 18 ετών, ακροτηριασμοί. χθε, για παράδειγμα, στην πόλη του Μασχάτ ακροτηριάστηκε ένας άνθρωπος ε, του έκοψαν τα χέρια. Ήταν ένα ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολύ συχνά δημοσιογράφοι, συνήγοροι, δικηγόροι αντιρρησίες ή αντιφρονούντες, ε, όσοι απλώς έχουν αντίθετη γνώμη από την κυβέρνηση κινδυνεύουν να συλληφθούν. Όσοι έχουν ε, κατηγορήσει την κυβέρνηση για νοθευμένες εκλογές υφίστανται ψυχολογικές διώξεις, ε, σωματικές, απειλές κατά της σωματικής και ψυχικής τους υγείας γίνονται τεράστιες ε, διακρίσεις, πολλές φορές εις βάρος των γυναικών, εις βάρος ε, φιλετικών ή θρησκευτικών μειονοτήτων. Δυστυχώς στο Ιράν εξακολουθούμε να έχουμε αυτή την ε, βάναυση και ε, μεταχείριση των γυναικών που μερικές φορές είναι σαν να είναι σκλάβες, το ίδιο και τα παιδιά που υφίστανται κακοποίηση πολύ συχνά. Δυστυχώς γίνεται φιλτράρισμα των, πολλών ε, δικτύων πληροφορικής, μπλοκάρονται δορυφορικές ε, αναμεταδόσεις. Είναι κατάφορη η παραβίαση της προσωπικής ελευθερίας στο Ιράν. Είναι τραγικά αυτά τα φαινόμενα και δείχνουν πόσο επισφαλής είναι η θέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Σήμερα λοιπόν είναι σημαντικό να δείξουμε ότι μας ενδιαφέρει αυτή η χώρα και ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε σε χώρες που καταστρατηγούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη ζωή όπως το Ιράν να χρησιμοποιούν διάφορα προσχήματα και μέσω νομοθετικών διατάξεων ή μέσω του νόμου της Σαρία να παραβιάζουν κατάφορα τα δικαιώματα των πολιτών τους. Έχουμε δύο είδη παράβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Το ένα αφορά το, την εθνική νομοθεσία και το εθνικό δίκαιο του Ιράν και δεύτερος λόγος είναι η εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων ε, ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάντως, ελπίζω ότι οι δυτικές χώρες θα καταφέρουν να ορθώσουν το παράστημά τους απέναντι σε αυτούς που καταστρατηγούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω ότι οι δυτικές δυνάμεις, οι δυτικές χώρες μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο και να μας βοηθήσουν ε, να προασπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι είναι καθήκον όλων μας να τεθεί ένα τέρμα σε αυτές τις παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι είναι προς το πολιτικό συμφέρον όλων μας, ακόμη και των δικών σας χωρών. Εγώ ε, γεννήθηκα και έζησα σε μια χώρα όπου καθημερινά παρατηρούμε κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και δεν είναι μόνο οι δυτικέ χώρε, αλλά οποιαδήποτε χώρα του κόσμου που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να συνεργαστεί με τι υπόλοιπε για να βοηθήσουμε τα θύματα αυτών των παραβιάσεων. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και αυτό το ζήτημα. Τα θύματα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ πιο σοβαρό ζήτημα, ακόμη και από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και αν μια χώρα καταστρατηγεί τα δικαιώματα των ίδιων της των πολιτών, των ίδιων της των υπηκών, σημαίνει ότι δεν πρόκειται να σεβαστεί κανένα δικαίωμα ούτε άλλης χώρας. Οπότε αν μια τέτοια χώρα έχει στρατιωτική ισχύ και τη χρησιμοποιήσει να διαπράξει και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Γι' αυτό θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εστιάσουμε την προσοχή μας στα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί η στάση μιας χώρας στο θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων λέει πολλά για την ίδια τη χώρα και σχετίζεται και με το πυρηνικό θέμα. Πιστεύω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να βρεθούν ως ύψη προτεραιότητα στο πρόγραμμα όλων των χωρών. θα πρέπει να βοηθήσουμε τον Ιρανικό λαό, για παράδειγμα, να έχει πρόσβαση στο Ιντερνετ, απρόσκοπτη πρόσβαση στο Ιντερνετ, ή να αφυπνίσουμε τον κόσμο προκειμένου να αναχαιτιστεί η λογοκρισία και τα προβλήματα στις ε, δορυφορικές αναμεταδόσεις. Επίσης, να φροντίσουμε, να ζητήσουμε να αποφυλακιστούν οι αντιφρονούντες Θα ήθελα να σας απευθύνω θερμή έκκληση να βοηθήσετε τους Ιρανούς που ζητούν άσυλο στις χώρες σας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ελεύθεροι στην πατρίδα τους και έχουν προσφύγει σε εσά ζητώντας μια προστασία και το άσυλο. Παρακαλώ μην τους κόψετε το δρόμο, διευκολύνετε, διευκολύνετε τους να λάβουν άσυλο. Ε, καλό θα ήταν να οργανωθούν και εξεταστικέ των πραγμάτων επιτροπέ. Για παράδειγμα, ο κύριο Αχματινιτζάντ είπε στη Νέα Υόρκη ότι θα πρέπει να γίνει μια εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή για την 10η Σεπτεμβρίου. Γιατί να μην ζητήσετε κι εσεί τέτοια ε, εξεταστική επιτροπή για το Ιράν ή ακόμη και διεθνέ δικαστήριο για το Ιράν. Και θα πρέπει να προσελκύσετε και την υποστήριξη άλλων ε, Ισλαμικών χωρών αλλά αντίστοιχο λόμπι κάνει ο Αχμαντινετζάτ. Είδατε τι έκανε στο Λίβανο. Πριν πάει στο Λίβανο, έδωσε 350 εκατομμύρια δολάρια, δόρισε 350 εκατομμύρια δολάρια στη λιβανική κυβέρνηση για να κερδίσει την υποστήριξή της. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη δήλωσή σας κύριε Ψαφάη. Είναι μια σημαντική μαρτυρία ε, να στείλει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία αποστολή για να αυτή την κατάσταση τόπου. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σάρπ και μετά στην κυρία Οτμελέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον κύριο Μαχαμαντή για την τόσο έντονη αυτή δήλωση που έκανε. Θα ήθελα να σας υποβάλω κάποιες σημαντικές ερωτήσεις το τι μπορεί να κάνει δηλαδή κάνουμε εμείς για να βοηθήσουμε τους ε, Ιρανούς. Ο πρόεδρος Ομπάμα ε, προετοίμασε μια εκτελεστική ε, διαταγή για να βοηθήσει παραδείγματος χάρη να φορούσε αυτό 27 άτομα. Αυτό βοηθάει. Ε, είπατε τι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι ο ρόλο κατά γνώμη τη Τουρκία όλα αυτά αν ξέρετε κάτι, γιατί πολλοί φεύγουν από το Ιράν και πάμε στην Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έντονη σχέση με την Τουρκία και δεν ξέρω αν βλέπετε να υπάρχει μία, ένας τρόπο ε, τρόπος συνεργασίας με την Τουρκία ενώ των Ιρανών. Ή αναφέρθηκα στην ανάγκη χορήγησης ασύλου. Αν έχετε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα θα ήταν καλό. Έχουμε το πρόγραμμα των ε, των πόλεων προσφυγή ε, city shelter όπως τα λέμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ακόμα λειτουργικό αλλά θα γίνει λειτουργικό όσον αφορά του ζητούν άσυλο στην ε, Τουρκία. Δεν ξέρω κατά πόσον γνωρίζετε πόσο καλά λειτουργεί ε, η Επιτροπή του, Ευρωπαϊ... Εθνών ε, για, τα... για τους πρόσφυγες Αυτά. Έχω και άλλε ερωτήσει, αλλά ίσω και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι να μπορούν να υποβάλουν κάποιε παρόμοιε ερωτήσει. Ευχαριστώ. Πρώτα, ευχαριστώ κύριε Σάκερ. Θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι σήμερα λαμβάνει η χώρα μια στάντσα ενταξία ενό σημαντικού δικτύου αυτών των, ε, των πόλων καταφυγίων και είναι πάρα πολύ καλή λοιπόν η παρατηρήσή σας, πάρα πολύ επίοξη. Η κυρία Σότμιλε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα αναφερθώ μόνο στην αρνητική ποινή. Και άλλες ερωτήσεις είναι σημαντικές, αλλά εγώ θα βρεθώ σε αυτό. Από ό,τι κατάλαβα υπάρχει νομοσχέδιο στην ε, Ιραντική ε, Βουλή που υποβλήθηκε το 2000 Τρία, για να καταργηθεί ο λιθοβολισμός. Και υπάρχει γιατί πολλοί προσπέσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Ιράν τη ζήτησαν. Αλλά προφανώς τώρα μπλοκάρεται αυτό το νομοσχέδιο και θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσον υπάρχει καμία πιθανότητα να επανυποβληθεί και το νομοσχέδιο αυτό και να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την αποστολή αυτή, είναι κάτι που βέβαια το, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους ε, εισηγητές και νομίζω ότι δεν έχει το θέμα καμία συγκεκριμένη άδεια επίσκεψη και υπάρχει εδώ μια αντίφαση γιατί έχουμε μια αντιπροσωπεία του Ιράν που θέλει να πάει εκεί Τώρα μας είπαν όμως ότι μπορούμε να πάμε μόνο εφόσον η κυρία Στιάνη δεν είναι πια αντιμετωπή με την θανατική ποινή. Και θα πρέπει να το δούμε αυτό. Δηλαδή, ή θα είναι αυτή μια πολιτική φίλου, δεν μπορούμε να πάμε ούτε στη Σαουδική Αραβία, στη ΣΥΠΑ ή στην Κίνα, ή θα δούμε τι θα κάνουμε να είμαστε πιο σοβαροί. Βλέπω εδώ την Κομισιόν, του κύριο Μουσίνη. Είναι ότι έχει καλά νέα. Θα έχουμε την εκπομπή Euronews στη Φαρσή. Τέλειο Οκτωβρίου νομίζω. Δεν ξέρω κατά πώς θα μπορέσουν να επιδράσουμε στο πρόγραμμα αυτό αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ε, τα στοιχεία αυτά παραδείγματος για την κατά, ε, κατάληξη ποινής γιατί στο ιστορικό του Ιράν οι πολίτες δεν ξέρουν αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Χολμήρα. Λέει πρόεδρος. Αν ο κύριος Κουσίνη θέλει να πάρει το λόγο σύντομα θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής να του το δώσω. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε και για τα καλά λόγια της κυρίας Ροχπίλε. Η εκδοχή των Euronews σε φαρσί θα αρχίσει να εκπέμπεται σε μερικές μέρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευρύνουμε τις δυνατότητες. Οι Ιρανοί τηλεθεατές να μπορούν να ξέρουν τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό το πρόγραμμα θα αρχίσει νομίζω τέλη του μηνός αυτού ή ίσως στην ε, αρχές του επόμενου μήνα. Και συμπεριλαμβάνονται δύο πράγματα. Καταρχήν, δεν είναι καινούριο κανάλι που δημιουργείται. Είναι αυτή η μορφή του γεωρονιούς που υπάρχει. Θα προσθεθεί απλώς η γλώσσα φαρση στις άλλες γλώσσες που συμπεριλαμβάνουν αραβικά, ρωσικά και τουρκικά. Το δεύτερο είναι ότι εμείς θέλαμε, δημιουργώντα αυτή τη δυνατότητα, να στοχεύσουμε στην δυνατότητα να μας δουν για να μας ακούσουν περισσόφωνοι ανά τον κόσμο. Δηλαδή όχι μόνο στο Ιράν που είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικό αλλά στις γειτονικέ χώρες υπάρχουν σημαντικές κοινότητες που μιλούν την ελληνική γλώσσα, μια διασπορά πάρα πολύ σημαντική ανά τον κόσμο. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί η Euronews έχει ολόκληρο στόλο δορυφών που μπορεί πραγματικά να εκπέμψει παντού. Κατά τα άλλα, σας ζητώ συγγνώμη που άργησα. Από την άλλη μεριά άκουσα με, προσοχή τα μηνύματα του κυρίου Μουσταφάη. Καταρχήν να σα πω ότι προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διπλωματικά κανάλια που έχουμε στη διάθεσή μα για να αποστείλουμε πολύ ξεκάθαρα μηνύματα στι ιρανικές αρχέ. όσον αφορά τι ανησυχίε με δηλαδή, τόσο δύσκολη κατάσταση εδώ και πάνω στη χώρα αυτή. Και δεύτερον, οι Ιρανικές αρχέ, η Ιρανική κυβέρνηση θα πρέπει να σέβεται τι διεθνεί υποχρεώσει που έχει αναλάβει υπογράφοντα και επικαιρώνοντα μια σειρά συμβάσεων, παραδείγματο κατά την προστασία ανθρωπών για τι βασικέ ελευθερίε, ε, τι πολιτικέ ελευθερίε κλπ. Υπενθυμίζοντα τι υποχρεώσει του, δεν ε, θέλουμε να δίνουμε την εντύπωση ότι παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά της ε, χώρας αυτής Απλώς πρόκειται για κάτι που ελεύθερα έκαναν ε, αβίαστα οι Ιρανοί, υπέγραψαν δηλαδή αυτές τις βάσεις και τώρα είναι δίκαιο να το ζητήσουν μια που τις υπέγραψαν να τις σεβαστούν τις διεθνείς αυτές τις βάσεις. Ε, εκτός αυτού θα ήθελα να υπενθυμίσω διάφορες δηλώσεις που έκανε η πατή εκπρόσωπος η Καθρινάσον, φέτος. Δέκα δηλώσεις, ε, διάφορες ε, διατυπώσει που κάναμε στη Τεχεράνη και στις Βρυξέλλες, διάφορα διαβήματα που προσπαθήσαμε να οδηγήσουν σε λογικές και σημαντικές συζητήσεις με τις Ιρανικές αρχές, πιστεύοντας την προσοχή τους στη γενική κατάσταση και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά που ακούσαμε στο διαδίκτυο, στα κινητά τηλέφωνα, στις ε, επικοινωνίες με δορυφόρο. Υπάρχει μια έντονη συζήτηση με τις Κομισιόν Συμβουλίου Κρατών Μελών και εμπειρογνωμόνων και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ελπίζω βάσει όλων αυτών των μελετών να μπορέσουμε να καταστήσουμε την παρέμβασή μας πιο αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Πρώτα σας ευχαριστώ για τα τόσο ενδιαφέροντα και ενημερωτικά που μας είπατε και Λουσίνη ίσως η άρμαδη υπηρεσία του Κοινοβουλίου θα μπορούσε να έχει κάποια συζήτηση με την Euronews πώς αυτή η πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να τονιστεί καλύτερα στα προγράμματα Euronews, στις διάφορες γλώσσες αυτές. Επίσης θα ήθελα να σας πω κύριε Πουσίλη, ότι πήραμε σήμερα μία γραπτή, θα πάρετε μία γραπτή ερώτηση σήμερα από κύριο Σάρκη και την υποφαινόμενη για το τι πρόκειται να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μπορεί να κάνει όσον αφορά αυτά τα ε, πρότυπα τηλεπικοινωνίας και τι μπορεί να γίνει ε, όταν τα μέσα αυτά χρησιμοποιούν για τον έλεγχο των πολιτών. Τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριο Σέμχια, αντιπρόεδρο σε αυτή την σειρά, σε αυτό το γύρο συνεδρίσεων. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μουσταφέη. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να κάνουμε κάποια σκέψη και μετά να θέσω και μία ερώτηση. Όντως, το Ιράν είναι μια χώρα που καταστρατηγεί μαζικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατάφορα και μερικέ φορέ έχει και επιδεικτικό χαρακτήρα αυτή η καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για, το, για παράδειγμα, τρόπος εκτέλεσης τη θανατική ποινή. Άλλο παράδειγμα είναι η δίωξη της αντιπολίτευσης μετά τις τελευταίες προεδρικές εκλογές. Βέβαια, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το Ιράν με την κατάσταση άλλων χωρών. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το Ιράν με τη Βόρεια Κορέα, που είναι τελείως απομονωμένη χώρα. Στις τελευταίες προεδρικές εκλογές τουλάχιστον είχαμε πολλούς υποψήφιους στο Ιράν, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί. Και για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα είχαμε τόσο έντονη αντιπολιτευτική δραστηριότητα. Μετά τη σκέψη αυτή θα ήθελα να σας κάνω και μία ερώτηση. Εσείς πώς εκτιμάτε, πώς αξιολογείτε την στάση που παρατηρούνται στο Ιράν. Γιατί μιλούμε πολλές φορές για το παρόν, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε την παρούσα κατάσταση σε μια εξελικτική διαδικασία και με κάποια προοπτική. Η κατάσταση σήμερα στο Ιράν είναι καλύτερη, γιατί οι πρόσφατες προεδρικές εκλογές ήταν, συγκλώνησαν αρκετά, πιστεύω, το Ιράν. Μετά τις τελευταίες προεδρικές εκλογές, εκλογές. Βλέπετε μία τάση του Ιράν για περισσότερη ε, εφαρμογή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ή μήπω εξαιτία τη ε, ενίσχυση τη αντιπολίτευση οι Ιρανικέ αρχέ εξωθούνται σε μεγαλύτερο ριζοσπαστισμό και σε πιο αυστηρή και ανελαίτη δίωξη. Πώς ε, διορθώνουν την πολιτική τους οι ιρανικέ αρχές με βάση τι τελευταίε εξέλιξεις. αυτέ τι τάσει θα ήθελα να μα περιγράψετε. Και τώρα θα επιστρέψουμε στον κύριο Μουσταφά για πέντε λεπτά για να μας απαντήσει σε ερωτήσεις που ακούστηκαν από τα μέλη της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά και πάλι για το ότι δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όσους ε, μίλησαν για την κατάσταση στο Ιράν. Μετά τις Ιρανικές εκλογές διαπιστώσαμε ότι μεγάλος αριθμός Ιρανών κατέβηκαν στους δρόμους για διαμαρτυρία και είχαμε πραγματικά μαζικά συλλαλητήρια και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Βέβαια, σε αντίθεση με άλλες χώρες, το Ιράν Η... Ο μεγάλος πλούτος της χώρας οφείλεται στα κοιτάσματά της σε πετρέλαιο και στους φυσικούς της πόρους γενικώ. Και εξαιτία της ισχύω που λαμβάνει το Ιράν, που λαμβάνουν οι Ιρανικές αρχές από το φυσικό πόρο και από το πετρέλαιο, μπορεί να καταπιέσει τον λαό. Χάρη στον πλούτο που συσσωρεύει, το Ιράν προσλαμβάνει περισσότερους αστυνομικούς, ενισχύει τις στρατιωτικές δυνάμεις και άρα και τον κατασταλτικό της μηχανισμό. Ο πλούτος δηλαδή της ε, χώρας αυτής χρησιμοποιείται για την ε, ενίσχυση της αστυνομίας, για τον έλεγχο και την καταστολή του λαού. Επίσης, χάρη στον πλούτο που έχει η χώρα αυτή, αγοράζει η τεχνολογία και τη χρησιμοποιεί. Οχτώ άνθρωποι που ήταν από τους βασικούς παραβιαστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων τιμωρήθηκαν από τον πρόεδρο Ομπάμα και αυτή ήταν μια πολύ σημαντική πρόοδος και είχε πολύ θετικό αντίκτυπο στο Ιράν. Παρόμοια διαβήματα θα μπορούσαν να γίνουν και κατά άλλων παραβατών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι διαπραγματεύσει με το Ιράν συνεχίζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πολλέ συμβάσει και συνθήκε έχουν εγκριθεί από το Ιράν, όπω η συνθήκη για το σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών. Παρά την επικύρωση όμω αυτή τη συνθήκη, βλέπουμε ότι εξακολουθούν να γίνονται εκτελέσει ανηλίκων στο Ιράν. Το Ιράν έχει πολλέ προκλήσει να αντιμετωπίσει και προσπαθεί να χρησιμοποιήσει και νέε μεθόδου. Αλλά δυστυχώ η μέθοδοι αυτή είναι καταπιεστικές και κατασταλτικές. Πέρυσι συμπεριλήφθηκε στην ειρηνική νομοθεσία δυνατότητα καταδίκηση σε θανατική ποινή ακόμη και bloggers. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας στο ΙΕ θα πρέπει αντί να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις που σε τελική ανάλυση πλήττουν τον ε, Ιρανικό λαό, να επιβάλλει πολιτικές κυρώσεις, γιατί οι πολιτικές κυρώσεις ουδέποτε δεν επιβλήθηκαν εις βάρος του Ιράν. Οι ηγέτες του Ιράν είναι αυτοί που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτοί ελεύθερα κινούν, διακινούνται στον κόσμο, πηγαίνουν στο εξωτερικό και εκφωνούν ελεύθερα ομιλίες και χρησιμοποιούν ουσιαστικά άλλες χώρες προκειμένου να ανοίγουν ε, λογαριασμούς σε αλλοδαπό συνάλλαγμα και όλα αυτά γίνονται ανενόχλητα από τους ηγέτες της Ιρανικής ηγεσίας, της Ιρανικής κυβέρνησης σε αντίθεση με το λαό που καταπιέζεται από τις οικονομικές κυρώσεις. Πολιτικές κυρώσεις λοιπόν χρειάζονται πρώτα απ' όλες βάρος του Ιράν. Αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να γίνεται επέμβαση στην εσωτερική πολιτική του Ιράν. Η κοινωνία μας όμως έχει πια γίνει παγκοσμιοποιημένη. Δεν μπορούμε να μένουμε αδιάφοροι για αυτά που συμβαίνουν στο εσωτερικό του Ιράν. Όλες οι χώρες θα πρέπει να ελευθερωθούνται. Και η Βόρεια Κορέα χρειάζεται την υποστήριξή μας. Και οι Κινέζοι χρειάζονται την υποστήριξή μας. Και οι Ιρανοί. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να γίνει προτεραιότητα. Να αφήσουμε κατά μέρο το συμφέρον, να καθίσουμε από κοινού και να αναζητήσουμε κοινέ λύσεις και τους κατάλληλου μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Thank you so much, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε που ήρθατε να μιλήσετε ενώπιον μας και σίγουρα θα έρθουν σε επαφή μαζί σας βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μελλοντικά. Νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε αυτό το θέμα των κυρώσεων και περιορισμών στα ταξίδια. Ε, από διάφορες χώρες όπου υπάρχουν σοβαρότατες παραβιάσεις ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, σίγουρα δεν πρέπει να επιτρέψουμε την ελεύθερη μετακίνηση αυτών των ανθρώπων. τώρα, έχουμε ακόμη τρία τέταρτα, θα αφιερώσουμε στην τροποποίηση του κανονισμού για τον Frontex, τροποποίηση λοιπόν του κανονισμού του Συμβουλίου που γίνεται τώρα. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων μας έδωσε την άδεια έδωσε την ε, άδεια στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να γνωμοδοτήσει επί του θέματος και η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αναλάβει την σύνταξη της νομοδότης τελική. Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για την 1η Δεκεμβρίου στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Η κυρία Λόχ Μπίλερ είναι η συγγήτριά μας, η συντάκτρια μάλλον της νομοδότησης. Ε, να σας υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα που είναι ενδεικτικό. Σήμερα πρώτη εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης κυρίας Λοχμπίλερ. Η προθεσμία υποβολή τροπολογιών για το σχέδιο αυτό προτείνεται ε, να οριστεί στις 25 ε, Οκτωβρίου μέχρι τις 12. Στις 29 Νοεμβρίου θα γίνει δεύτερη εξέταση στην υποεπιτροπή μας και εξέταση των τροπολογιών του σχεδίου και ψηφοφορία, είπαμε, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποδέσεων την 1η Δεκεμβρίου. Τέλος, η Επιτροπή, ε, ε, η καθήλυνα αρμόδια, δηλαδή η Επιτροπή ε, Ελευθεριών, θα ψηφίσει στις 9 Δεκεμβρίου του 2010 να σας εξηγήσω ποιοι είναι παρόντες για να σχολιάσουν ε, το σχέδιο γνωμοδότης και το σχέδιο τροποποίησης του κανονισμού. Νίκολας Λεζέρ, ε, Διευθυντής ε, ε, του, της, ε, του Ευρωπαϊκού Γραφείου της ε, Διεθνούς Αμνηστίας, ο κ. Κριστάφ Κίσλερ, που είναι βαθμός αξιωματούχος της υπηρεσίας μεταναστών στην Ευρώπη και η κυρία Μάντλιν Γκάρλικ, επικεφαλής του τμήματος πολιτικής του, της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΗΕ και συγκεκριμένα του γραφείου της στις Βρυξέλλες. Ε, ο Frontex εκπροσωπείται από τον κύριο Ρίτσαρντ Άρες Μπάμκαρ. Η συντάκτρια η κυρία Λόχ Μπίλτερ θα μας παρουσιάσει τώρα το σχέδιο γνωμοδότησης. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω γράψει η αιτιολογική έκθεση και τις τροπολογίες που έχετε μπροστά σας. Δεν πρόκειται να αναφερθώ μία προς μία, θα σας δώσω μια γενική εικόνα Ποιε είναι αυτέ οι προτάσει εμεί ως Επιτροπή Ανθρωπινών Δικαιωμάτων διαφωνόμαστε ιδιαίτερα για το ότι το πλαίσιο εργασία του Frontex θα πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα και επίση θα πρέπει ε, σωστά να εφαρμόζονται καθ' όλη τη διάρκεια τη εργασία του Frontex. αναφέρεται ότι θα πρέπει οπωσδήποτε η Frontex να εκτελέσει το έργο της και να λάβει υπόψη αυτές τις πτυχές. Ξέρουμε και μέσα στα πλαίσια του κοινοβουλικού πλαισίου γνωρίζουμε τα φρικτά που διαμείβονται κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα Frontex, υπάρχουν διαφορετικά συστήματα εξασφάλισης των σύνορων και όλα θα πρέπει αυτά να ενταχθούν σε μια γενική εικόνα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ε, μετανάστευση και την χορήγηση δικαιωμάτων ασύλου. Εμείς θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας καταρχήν στην Frontex. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω όμως τις στήσεις που είχαμε μέχρι στιγμής. Ήμουν και τμήμα μια που προκάνωσε η Επιτροπή Λίμπε στη Βαρσοβία πριν από δύο στην ε, έδρα του Frontex και εκεί συζητούνται διάφορε οδηγίε που είναι εκτός ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραδείγματο χάρη, ποια είναι η δυνατότητα επιβολή δικαιωμάτων από τι εθνικές ε, ε αρχές, αρχές σε σχέση με την Frontex. Πόσα χρήματα θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έχουμε τώρα ένα πάρα πολύ σημαντικό προπελαιό στη Frontex και κατά πόσο θα αυξηθεί ή αν επαρκεί. Επίσης στην Βαρσοβία, μια που μου λένε ε, οι επικεφαλής του Frontex που χρειαζόνται περισσότερη διαφάνεια, είπα ότι ωραία, έχουμε αυτή την ακρόαση και θα την κάνουμε να έρθει και κάποιος από τη Frontex. και θα πρέπει ίσως και στο μέλλον να είναι δεσμευτική αυτή η παρουσία, να έχουμε συνεχή παρουσίαση της σωστής εφαρμογής των ε, διατάξεων Frontex και της εργασίας του Frontex. Λοιπόν, στην ιδεολογική μου έκθεση τονίζω ότι αυτό που έχει κάνει ήδη η Κομισιόν και έχει πει η Κομισιόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ καλό βασικό η εργασία του Frontex να ακολουθεί πάντα τις αρχές προστασίας των δικαιωμάτων. Έχουμε μια νέα κατάσταση μετά την συνθήκη της Λισαβόνας που δημιουργεί ένα νέο νομικό πλαίσιο όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να, ε, ανισχυθ, να λάβουν πόσο ότι ενισχύεται η εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. όσον αφορά τη διεύρυνση εντολής αναφέρεται ότι εξετάζουμε ότι όταν η Frontex διευρύνει την αρμοδιότητές τη, ε, θα πρέπει να παρακολουθούμε εμείς να σέβονται παρόλα αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα, μια που πρόκειται για μια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην τα λέμε αυτά δηλαδή γενικά και αόριστα, αλλά να φροντίσουμε να ε, προστατευτούν, εγγυηθούν και να προωθηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι μια ιδέα που διέπει όλες αυτές τις ε, προτάσεις. Εισαγωγικά. Έχω να σας πω ότι τόνισα ότι υπάρχουν ορισμένα πολύπλοκα θέματα που αφορούν το δίκαιο των εθνών, παραδείγματος χάρη, όσον αφορά την διάθεση ναυαγών. Είχαμε στα πλαίσια της ομάδας των Πρασίνων μία ακρόαση και με προσώπους της Κομισιόν πυρογνώμονες νομικών θεμάτων που δεν μπορούσαν να μας δώσουν μια ξεκάθαρη παρουσίαση και εγώ στην ε, έκθεσή μου λέω ότι θα πρέπει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να ασχοληθεί με τη διαλεύκανση αυτού του σημαντικού σημείου. Λοιπόν, καταρχήν χαιρετίζουμε τις προτάσεις Κομισιόν. Κατόπιν ε, υποβάλλουμε συγκεκριμένες ε, απαιτήσεις που λένε ξεκάθαρα πώς θα εργαστούμε σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταρχήν είναι αξιολόγηση της δραστηριότητα ε, της ε, υπηρεσία αυτή Frontex. Το ζήτησε ήδη το 2008 το κοινοβούλιο αυτό. Να υπάρχει δηλαδή μια ανεξάρτητη αξιολόγηση και στο αίτημα αυτό του κοινοβουλίου δεν υπήρξε καμία αντι... Ε, αντίδραση. Θα πρέπει τώρα να ζητήσουμε εσωτερική και εξωτερική ε, αξιολόγηση συνολική και ανεξάρτητη που να περιλαμβάνει και τους φορείς που συνεργάζονται με τον Frontex όπως τον Οργανισμό για Θεμελιώδη Δικαιώματα και τις αρμόδιες ε, μη κυβερνικές οργανώσεις. Και όσον αφορά την αξιολόγηση αυτή αναφερόμαστε σε πενταετία. Εγώ όμως θα ήθελα να γίνεται αυτό ετησίως μια που θα πρέπει να υπάρχει και ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Frontex. Περαιτέρω, συστήνω να μην αναφέρεται μόνο όπως λέγεται τώρα ότι η εξολόγηση θα πρέπει να αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και γενικά, αλλά θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Να πούμε, θα πρέπει να αναφέρεται ακριβώς τι γίνεται και κατά πόσον τηρείται η χάρτα. Επίσης λέμε ότι χρειαζόμαστε μια εποπτεία ανεξάρτητη για την τήρηση αυτών των ε, υποχρεώσεων. όχι μόνο αν ε, προωθούνται οι στόχοι αλλά και αν πληρούνται τελικά στην πράξη. Και γι' αυτό είναι καλό να διευρυνθεί η συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΕ για τους πρόσφυγες, ούτως ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στην προετοιμασία και την εφαρμογή όλων των κοινών επιχειρήσεων, ιδίως όταν πρόκειται για θέματα που σχετίζονται με το άσυλο. Αυτό που είναι καινούριο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει αναφορά περιστατικών αυτό συγκεκριμένο περιστατικό φαίνεται ότι είναι βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο θα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιον τρόπο ούτω ώστε να μπορούμε να ξέρουμε ποιο είναι υπεύθυνο για ενδεχομένε καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια άλλη πρόταση είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν τακτικές εκπαιδεύσει για τους συνεργάτες της Frontex και αυτό σε συνεργασία με, με την Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αυτό είναι σημαντικό και επίσης συνεργασία μη κυβερνητών οργανώσεων και για την ε, προετοιμασία των προγραμμάτων ε, ε, κατάρτισης και όσον αφορά την πραγματοποίησή τους. Θα πρέπει να υπάρχει μία ομάδα υπερογνωμόνων στους οποίους θα πρέπει να έχει πρόσβαση η Frontex που να γνωρίζουν τη διεθνή προστασία συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων ε, προστασίας των ετούντων άσυλο που θα γνωρίζονται επίσης και τα θέματα της διεθνούς προστασίας ιδιαίτερα εκείνων που έχουν περισσότερη ανάγκη προστασίας. Έχουμε εδώ τους εμπειρογνώμονες που θα αναφερθούν στις λεπταμέρειες. θα αναφερθώ περισσότερο. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες και όλους όσους θα πάρουν το λόγο. Ήμουν πάρα πολύ ευγνώμων για τις ε, λεπτομερείς προτάσεις και γνώσεις που διέθεσαν στο Κοινοβούλιο. Από την Επιτροπή ΛΥΜΕ δεν έχω ακόμα ακούσει πώς ε, λαμβάνουν υπόψη οι τροπολογίες μας. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να είναι ενήμερο μπορούσε να βελτιωθεί, να είναι πιο ευρία δηλαδή αυτή η ενημέρωση. Και υπήρχε και μια, ένας διάλογος, αν θέλετε, μεταξύ ΛΥΠΕ και του Ευρωπαϊκού Αρμοδίου για την Προστασία των Δεδομένων. Δεν ξέρω το αποτέλεσμα της επαφής αυτής, αλλά οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντικό να προετοιμάσει μια πολιτική προστασία των δεδομένων Frontex. Γιατί όταν εγώ στη Βαρσοβία ρώτησα τι γίνεται με την πρόθεση και των στοιχείων των ατόμων που περνάνε από τις υπηρεσίες του Frontex, και μου είπαν ότι δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη πολιτική. Αν δεν υπάρχει όμως καμία πολιτική και αν δεν τηρούν αυτά τα στοιχεία, πώς θα μπορέσουμε να ελέγξουμε ως βουλευτέ. Ωραία. Αυτά εισαγωγικά από μένα. Thank Σας ευχαριστούμε κύριε Λόχμπίλερ. Όπως είπατε, είχαμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προσπαθεί να περιλάβει περισσότερα πτυχέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κανονισμό. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στο σκιώδη εισηγητή, τον κύριο Κουδουτσάκο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κυρία Πρόεδρε, είναι χαρά μου που έχω τη δυνατότητα να συμμετέχω στην εργασία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ερχόμενο από την ΑΦΕΤ, αλλά και, αν μου επιτρέπετε να πω, από μια χώρα, την Ελλάδα, που είναι σήμερα η μοναδική πύλη μαζικών εισόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην οποία το δεύτερο τρίμηνο του 2010, το δεύτερο τρίμηνο του 2010, ε, πέρασε από τα σύνορά της το 90% του συνολικού αριθμού ε, των ε, συνανθρώπων μας που αποπειράθηκαν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετέχω εδώ για να συζητήσουμε σε μια πρώτη και γενική ανάγνωση, σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, το κρίσιμο θέμα της Frontex. Κύριε Πρόεδρε ε, και κύριοι συνάδελφοι, ο κοινός στόχος όλων μας είναι, πιστεύω, ένας αποτελεσματικός Frontex που θα ασκεί την αποστολή του με τον απαραίτητο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το στόχο αυτό υπηρετεί ικανοποιητικά η πρόταση κανονισμού που κατέθεσε η Επιτροπή. Η πρόταση αυτή δίνει έμφαση στην αρτιότερη προπαρασκευή, στον μεγαλύτερο συντονισμό και κατά συνέπεια στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση των επιχειρήσεων που αναλαμβάνει ο Frontex, χωρίς ταυτόχρονα, και αυτό είναι το σημαντικό, χωρίς ταυτόχρονα να επιτρέπει τον εκφυλισμό του σε έναν αυταρχικό μηχανισμό αστυνόμευσης και καταστολής. Συνεπώς, οφείλω να ομολογήσω ότι στην πρόταση κανονισμού η Επιτροπή επιτυγχάνει σε ικανοποιητικό ή ακόμα και σε μεγάλο βαθμό μια παραγωγική ισορροπία, μια δύσκολη και ευπαθή ισορροπία μεταξύ επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και ανθρωπιστικής ευαισθησίας και δικαιοσύνης. Οφείλουμε ε, λοιπόν και εμείς στη γνωμοδότησή μας να διαφυλάξουμε αυτή την ευπαθή ισορροπία και τόσο δύσκολο να επιτευχθεί. Ε, η πρόταση γνωμοδότησης συναδέλφου της κυρίας ε, Λουκ Μπίλερ έχει αναφυσβήτητα πολλά θετικά στοιχεία και την συγχαίρω για τη δουλειά που έχει κάνει. Ταυτόχρονα αισθάνομαι ότι πρέπει να πω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η πρότασή της κινείται προς την κατεύθυνση της ανατροπής αυτής της ευπαθούς και δύσκολης ισορροπίας για την οποία μόλις σας μίλησα. Παραδείγματο χάρη αυτό γίνεται όταν ε, υπάρχει η πρόθεση να εμπλακεί η, Frontex σε θέματα που εμφανώς βρίσκονται εκτός αρμοδιότητάς του, όπως παραδείγματο χάρη τα θέματα ασύλου Επίσης, όταν ε, υπάρχουν προτάσεις που, κατά την άποψή μας, ε, μερικές φορές επιβαρύνουν υπέρμετρα τις διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης, ε, διότι η πρόταση της συναδέλφου κινείται ορισμένες φορές πολύ περισσότερο και πολύ μακράν των ικανοποιητικών προβλέψεων που περιλαμβάνει ο κανονισμός της Επιτροπής ικανοποιητικών ρυθμίσεων που δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε. Παραδείγματο χάρη, στην πρόταση της Επιτροπής διευκρινίζεται το νομικό πλαίσιο τη ε, της Frontex και των επιχειρήσεών της, καθίσταται υποχρεωτική η καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενισχύονται αποφασιστικά οι δυνατότητες ελέγχου και διαφάνειας με τακτικές διαδικασίες αξιολόγησης και βεβαίως αναπτύσσεται ο κώδικας δεντολογία για τις περιπτώσεις επαναπατρισμού. Ε, επομένως, ε, βλέπουμε ότι ε, έχει επιτευχθεί αυτή η ισορροπία στην οποία σας είπα. Εμείς θα αντιμετωπίσουμε με ανοιχτό πνεύμα και με διάθεση συνεργασίας και συνεννόησης τις προτάσεις ε, της συναδέλφου κυρίας Λόγμπιλερ, έχοντας βεβαίως ταυτόχρονα σημειώσει τους προβληματισμούς τους οποίους σας ανέφερα. Με την ευκαιρία αυτή, κυρία Πρόεδρε, και χωρίς να θέλω να ε, παρατείνω περισσότερο από ό,τι είναι λογικό τη συζήτηση για τον κανονισμό της Frontex, θα μου επιτρέψετε, ελπίζω, να αναφερθώ επιγραμματικά και σε ορισμένα επιχειρησιακά ζητήματα ε, που αφορούν ε, την Frontex και τον κανονισμό. Παράδειγμα του χάρη, θεωρώ ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας της Frontex με τα κράτη-μέλη θα πρέπει προκειμένου να σταματήσει μια επιχείρηση να έχει προηγηθεί διαβούλευση και ενημέρωση της Frontex με τις φιλοξενούσες στην επιχείρηση χώρες. Κράτη-μέλη. Επίσης νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό και θα είναι δύσκολο να φανταστώ κάποιο επιχείρημα που θα πηγαίνει ε, αντίθετα από την ανάγκη διαβούλευσης, διαλόγου και τελικά ε, συναπόφασης μεταξύ Frontex και, φιλοξενού, και φιλοξενούσας ε, χώρας μέλους όταν ζητάμε ή όταν πρόκειται να συζητηθεί η εμπλοκή και η συμμετοχή στην επιχείρηση του Frontex τρίτης εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως χώρας. Ε, τέλος, ένα άλλο ζήτημα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να δούμε είναι κατά πόσον βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και είμαστε έτοιμοι να δούμε μια αξιολόγηση των εθνικών δομών δυνάμεων εξοπλισμού και πόρων που διαθέτουν τα κράτη-μέλη στον τομέα του ελέγχου των συνόρων, δηλαδή κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να δούμε έναν έλεγχο, να ασκείται έλεγχος από τη Frontex για θέματα που αφορούν το σκληρό πυρήνα εθνικής κυριαρχίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα ευρύτερο βεβαίως πολιτικό, αλλά πρέπει να μας απασχολήσει. Και τέλος, ε, εκτιμώ ότι είναι ασαφής ε, η προτινόμενη στον κανονισμό, στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής ασαφής η εισαγωγή του θεσμού των ανεξάρτητων συνοριοφυλάκων. Ε, πρέπει να δούμε τι ακριβώς αντιλαμβάνεται κανείς με αυτή την εισαγωγή του νέου αυτού θεσμού. Ε, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που με ακούσατε και προσβλέπω στη στενή συνεργασία με την ε, ε, κυρία Λόχ Μπίλερ που έχει το βαρύ καθήκον να φέρει σε πέρας αυτή την, αυτή την γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Ευχαριστούμε κύριε Κουμτσάκου, είστε στο σκιώδη ηγητής από το έλικο όπως είπαμε. Τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τους, που, από τους προσκεκλημένους μας να πάρουν το λόγο. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, δεν είναι και πρώτη φορά βέβαια, θα τα καταφέρουμε. Μπορείτε να είστε σύντομοι και να το χρόνο αγόρευσης να τον περιορίσετε σε 6-7 λεπτά, σίγουρα θα το καταφέρετε για να έχουμε χρόνο να ακούσουμε και τις αντιδράσεις των μελών. Ο κύριος Μεζέρα από τη Διεθνή Αμνηστία, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, μας δίνετε και πάλι την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την άποψή μας για αυτό τον τόσο σημαντικό κανονισμό. Μιλώ εξ ονόματος ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Μεταναστών και Εξορίστων και ε, εκ μέρους της Διεθνής Αμνηστίας. Ε, πολλοί άνθρωποι εδώ έχουν αξιολογήσει την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εξετάσει τα τεχνικά της σημεία. Ευχαριστούμε <clears throat> τους εισηγητές. Το σχέδιο πραγματικά οδεύει προς σωστή κατεύθυνση σε μεγάλο βαθμό και συμπεριλαμβάνει τα τα βασικά σημεία στα οποία θα αναφερθώ και εγώ σήμερα. Ε, τρία ε, πολύ θετικά στοιχεία υπάρχουν στην πρόταση. Πρώτον, διευκρίνηση του νομικού πλαισίου επιβεβαιώνεται ότι οι δραστηριότητες του Frontex υπάρχονται στον ε, τελωνιακό κώδικα Schengen και πρέπει να υλοποιούνται δυνάμει του κώδικα. Αυτός ο κώδικας ε, του Schengen ε, λαμβάνει υπόψη την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δικάζει κάθε διακριτική μεταχείριση, κατοχυρώνει την προστασία των ατόμων και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που υπάρχουν εχέγγυα για τις κοινέ επιχειρήσεις επιστροφής που προβλέπεται από τον τελωνιακό κώδικα, ούτως ώστε να γίνουν με ανθρώπινο τρόπο οι επιστροφέ αυτών των ανθρώπων και τέλο έμφαση που δίνεται στην κατάρτιση των συνοριοφυλάκων και άλλων στελεχών που συμμετέχουν σε επιχειρήσει ελέγχου των συνόρων. Καλωσορίζουμε αυτά τα πολύ θετικά βήματα που δέχουν προ τη σωστή κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά έχουμε διάφορε βασικέ ανησυχίε και ε, ε, υπάρχονται σε τέσσερι κατηγορίε. Πρώτον, νέο νομοθετικό πλαίσιο ε, που παραμένει πλήρω ασαφέ σχετικά με τη δράση που πρέπει να να λάβουν τα κράτη-μέλη και ο Frontex, ούτω ώστε να συμμορφωθούν με τι απαιτήσει του σχετικά με τα ανθρωπίνα δικαιώματα, παρότι προβλέπεται αυτό μέσα στο σχέδιο. Περιγραφή του νομικού πλαισίου, λοιπόν, και ε, διεξαγωγή των επιχειρήσεων, ούτω ώστε να προστατεύονται όλοι οι πολίτε, κυρίω τα ευπαθή άτομα, ε, φαρμακευτική, τεχνική αγωγή, νομική αρρωγή, πρόσβαση ε, σε διαδικασία αίτηση ασύλου, συγκεκριμένα μέτρα δηλαδή που περιγράφονται στην πρόταση, γιατί αλλιώς ε, θα παραμείνουν όλα αυτά καινού νόηματο και δεν θα γίνει σωστά η υλοποίηση. Δεύτερον, επέκταση των αρμοδιοτήτων του Frontex, ναι, αλλά η λογοδοσία, το πλαίσιο παραμένει ασαφές, ε, από τρεις πλευρές τουλάχιστον. Ε, λογοδοσία, λοιπόν λοιπόν δεν ε, ε, ενισχύεται ουσιαστικά ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπω θα έπρεπε μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνα, το Κοινοβούλιο δεν είναι σε καλύτερη θέση για να ενημερώνεται σωστότερα και να ασκεί τον εποπτικό ε, ρόλο του. Θα υποβάλλονται συστηματικά οι εκθέσει, αλλά δεν περιγράφει ο τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει συμμόρφωση με τι απαιτήσει. Δεν υπάρχει κανένα ρόλο για την κοινωνία των πολιτών και των ανεξαρτήτων παρατηρητών και στα πλαίσια του Frontex δεν υπάρχει διαβούλευση σχετικά με το πρόγραμμα εργασία, παράδειγμα παραδείγματο χάρη. Στην πράξη συνεχίζεται η διακυβερνητική διακυβέρνηση για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων ε, με μυστικοπάθεια και πλήρη έλλειψη διαφάνεια. Επίση, δεν υπάρχει απέτηση παρακολούθηση του Frontex για τι διαδικασίε ε, επαναπροώθηση, αντίθετα με τι ε, διαδικασίε επιστροφή. Ε, προβλέπεται μηχανισμό ε, καταγγελία περιστατικών, αλλά δεν είναι σαφές αν αυτό θα σχετίζεται με περιστατικά που συνιστούν παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρί. κατάλληλη παρακολούθηση. Δεν μπορούμε να κατοχυρώσουμε ότι θα ε, καταγράφονται, θα παρακολουθούνται τα συγκεκριμένα περιστατικά, ακόμη και στα πλαίσια των κοινών επιχειρήσεων επιστροφή Και τρίτον, η συνεργασία με τρίτε χώρε. ενισχύεται μεν, αλλά αυτό συμβαίνει χωρί να έχουμε συγκεκριμένε ρήτρε, δικλείδε ασφαλεία. Ε, έχουμε το σωστό πλαίσιο και πάλι, αλλά και πάλι δεν υπάρχει η σαφή περιγραφή των ειδικών μέτρων ε, με τα οποία θα μεριμνήσουμε ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα και να μην υπάρχουν παραβιάσεις. Ε, και τέταρτο και τελευταίο σημείο για ε, τις, τα θετικά ηχέγγια που υπάρχουν για τις κοινέ επιχειρήσεις επιστροφής ήθελα να πω ότι υπάρχει διπλασιασμός του αριθμού των περιπτώσεων 500% σε σχέση με προηγούμενα ποσοστά, οπότε ε, καλωσορίζουμε αυτά τα ηχέγγυα, αλλά υπάρχουν ελλείψεις και θα θέλαμε να γίνουν κάποιες προσθήκες. Ελπίζουμε αυτό να γίνει με οικοδομητικό τρόπο, παραδείγματο χάρη ε, ε, πρόσβαση χωρίς κόλλημα σε όλες τις εγκαταστάσεις του Frontex, οι κοινέ επιχειρήσει, τώρα που συνεργάζονται διάφορα κράτη-μέλη, αυτοί που εποπτεύουν πρέπει να μπορούν να δουν ε, την πορεία όλων αυτών που επιστρέφουν, ε, ούτω ώστε να μεριμνήσουμε ε, και να υλοποιείται σωστά η συμφωνία. Θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμό παρακολούθηση σχετικά με το τι συμβαίνει, παραδείγματο χάρη, όταν υπάρχει καταγγελία περιστατικού και στη συνέχεια έκθεση για τι Αποφάσει υποχρεωτικής επιστροφής θα πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση και μετά, όταν δηλαδή επιστρέψει ο λόγω άνθρωπος στην τρίτη χώρα. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπεζέρε. Ο κύριος Κέσλερ τώρα θα πάρει το λόγο για λίγα λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ έναν οργανισμό καθολικών που ασχολείται με τα θέματα των προσφύγων σε όλο τον κόσμο, προσφύγων και μεταναστών. Και θα ήθελα να σας κάνω κάποια σύντομα σχόλια ως προς τον κανονισμό Frontex. Η γραμματεία μου σύστησε να είμαι λακωνικός και περιεκτικός, γι' αυτό θα προσπαθήσω να μην επεκταθώ σε λεπτομέρειες. Θα ήθελα να σχολιάσω κάποιες λεπτομέρειες της γνωμοδότησης Λόχ Μπίλερ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που επισημαίνει η κυρία Λόχ Μπίλερ, ότι το θέμα των ε, χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιλαμβάνεται στη συνθήκη υποχρεώνει όλους τους οργανισμούς, ακόμη και τη Frontex, να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων και αυτών των μεταναστών. Και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτριστεί σε ένα λεπτομεριακό νομικό πλαίσιο που θα πρέπει να ισχύει για τον οργανισμό Frontex. Η Επιτροπή σας άκουσε σήμερα το πρωί, είτε άμεσα είτε έμεσα, τα, τους λόγους εξόδου από, μια, από την πατρίδα τους. Το ακούσαμε από τους αυτόχθονες πληθυσμούς, από τους εκπροσώπους τους, από τους εκπροσώπους του Ιράν και από εμπειρογνώμονες που μίλησαν για τη θανατική ποινή. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που οδηγούν τους ανθρώπους να φύγουν από την πατρίδα τους. Προσοχή λοιπόν. Όσοι φεύγουν για να γλιτώσουν από παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα ε, να τύχουν προστασίας. Θα ήθελα να επιστήσω την προστασία σας σε χώρες όπως η Λιβύη, το Μαρόκο, η Αλγερία που είναι χώρες διαμετακόμισης. Εμείς ε, συνεργαζόμαστε με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και βλέπουμε πολλές ανθρώπινες υποθέσεις όπου ακόμη και οι μετανάστες αυτοί αναγνωρίζονται παρόλο που αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες από τον ΟΗΕ δεν τη χάνουν τις στοιχειώδεις προστασίες και της ε, απόλαυσης ε, στοιχειωδών κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων. Μένουν εγκλωβισμένοι στις χώρες αυτές γιατί ούτε μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους ούτε μπορούν να προχωρήσουν στη χώρα προορισμού τους. Και πραγματικά μένουν εγκλωβισμένοι σε αυτήν την κατάσταση και δεν έχουν καμία δυνατότητα διεξόδου. Θα πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις χώρες αυτές που είναι χώρες διαμετακόμισης, διέλευσης μεταναστών και προσφύγων και την κατάσταση ιδιαίτερα στα σύνορά τους. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τις διατάξεις και τις τροπολογίες που πρότεινε η κυρία Λόχ Μπίλερ που εσχεί ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα που γίνεται το επίκεντρο της ανάλυσης και διέπουν και τις σχέσεις μας με τις χώρες. Ο εντοπισμός της ανάγκης προστασίας είναι σημαντικό θέμα. Η κυρία Λόχ Μπίλερ πρότεινε να δημιουργηθεί ένα πουλμι ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα επικουρούν το γραφείο του ΟΗΕ. Αξιόπινη αξιό, αξιέπαινε συγγνώμη αυτή η πρόταση, αλλά τι σημαίνει ακριβώς ε, ε, επικούρηση του γραφείου του ΙΕ για την εφαρμογή και ποιος θα είναι ο ρόλος αυτών των εμπειρογνωμόνων. Το γραφείο του ΙΕ έχει αντίστοιχη αρρωγή εμπειρογνωμόνων και σε άλλους τομείς θα πρέπει να έχουν και ρόλο παρατήρησης αλλά και λόγω στενή συνεργασία με αυτούς που δρούν σε δραστηριότητες διαχείρισης συνόρων. Συμφωνούμε με τις προτάσεις της κυρίας Λόχβιλερ, Αλλά το, εκεί που λέει άσυλο θα ήθελα να λέμε διεθνής προστασία γιατί η διεθνής προστασία είναι ευρύτερη, είναι και καλύπτει και την προστασία των προσφύγων, αλλά και την ε, προστασία των εκτοπιστέντων. Ενώ όταν λέμε άσυλο είναι πολύ πιο ε, συσταλτικός όρος. Προτιμούμε το άσυλο να το αντικαταστήσουμε από το διεθνής προστασία. Σε ό,τι αφορά την ε, καταγγελία ή την ε, αναφορά των περιστατικών, συμφωνούμε με την πρόταση για τις ε, για την ενημέρωση αυτή, αλλά αναφέρονται μόνο αξιόπιστες καταγγελίες. Ποιε όμως είναι οι αξιόπιστες καταγγελίε, ποιο θα κρίνει αν μια καταγγελία είναι αξιόπιστη. Δεν μπορούμε μόνο υπό, το, υπό τον όρο της αξιοπιστίας μιας καταγγελίας να ενεργοποιούμε την έρευνα μιας υπόθεσης, γιατί είναι πολύ αυθαίρετος αυτός ο χαρακτηρισμός. Κάποιες χώρες ήδη έχουν ξεκινήσει το θέμα της εποπτείας του ελέγχου των ροών επιστροφής. Συμφωνούμε με την τροπολογία της κυρίας Λόχμπίλερ για την παρακολούθηση αυτή, αλλά θα πρέπει να προσδιορίσετε στο κείμενο ότι ανεξάρτητη παρακολούθηση δεν σημαίνει ανεξαρτησία της Frontex, ανεξάρτητα από τη Frontex, αλλά ανεξάρτητα και από τις αρμόδιες αρχές των χωρών μελών. Αλλιώς θα υπάρξει πρόβλημα και σύγκρουση συμφερόντων. Αυτά ήταν ορισμένα σχόλια. Ελπίζω να ήταν αρκετά σύντομα και αρκετά περιεκτικά και να δώσουν και τροφή για περαιτέρω συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας κύριε Ήταν πολύ σημαντικές. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μάντλη Κάλλιν από το UNHCR, το Γραφείο των Βρυξελών. Ευχαριστούμε. Το γραφείο της ΥΠΑ της Αρμοσίας του Ιού επανειλημμένα ζήτησε ε, να υπάρχουν ηχέγγυα στην πολιτική μετανάστευση και διαχείριση των ιστορικών συνόρων για να υπάρχει προστασία και εύκολη πρόσβαση και ίσες ε, ε, δίκες μάλλον διαδικασίες απονομής ασύλου. Αυτό προβλέπεται από τις συνθήκες και η ΥΠΑ η Αρμοστία έχει συγκεκριμένο ρόλο παροχή συμβουλών στα κράτη-μέλη για αυτές τις διαδικασίες μεταξύ άλλων. Ε, βλέπουμε τις προτάσεις για το Frontex ε, που ε, έχουν άμεσες επιπτώσεις στους μετανάστες και, όσους, και στους ετούντες άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά δεν έχουμε συγκεκριμένη εντολή, υπάρχει όμως το κοινοτικό κεκτημένο και οι δραστηριότητες του Frontex πρέπει να συνάδουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα που προβλέπονται από το νομικό πλαίσιο μεταξύ των οποίων και παροχή ασύλου. Ε, σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής και την έκθεση της κυρίας Λόχμπιλερ προτείνουμε στον αναθεωρημένο κανονισμό να υπάρχουν ε, νέα εχέγγυα, δηλαδή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παροχή διεθνούς προστασίας. Μεταξύ αυτών να μας ε, καλωσορίζουμε την πρόταση περί ενίσχυσης ε, του νομικού πλαισίου. Δηλαδή ο οργανισμός αναφέρεται ρητά ότι πρέπει να δρά δυνάμει των διεθνών υποχρεώσεων. Επίσης υποχρέωση κατάρτισης του προσωπικού και των συνοριοφυλάκων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, σημαντικό βήμα και νέα νέα μέτρα σχετικά με τη διαδικασία επιστροφή. Η ύπατη αρμοστία συμφωνεί ότι η βασική πρόκληση για την τροποποίηση του κανονισμού είναι η πρακτική υλοποίηση, δηλαδή η τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά με τη διεθνή προστασία και μη επαναπροώθηση. Αυτά θα κατοχυρώνονται μόνο εάν οι επιχειρήσει επιστροφή αντανακλούν αυτέ τι απαιτήσει μέσω συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών προ του συνοριοφύλακες, είτε μιλάμε ε, για θαλάσσια, είτε σύν, αέρια σύνορα ε, και πρέπει να έχουν συγκεκριμένες οδηγίες και τα μέσα και τις απαιτούμενε δεξιότητες για να εντοπίζουν και να αντιδρούν σωστά στους ετούντες άσυλο. Αυτό αναγνωρίζοντας ε, το ότι το να αφήνουμε να εισέρχονται κάποιοι ετούντες άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέρος των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών της Frontex. Οπότε συστήνουμε πέρα από τις υφιστάμενες προτάσεις, δηλαδή καλύτερος προσδιορισμός του νομικού πλαισίου και συμπερίληψη σαφέστατων υποχρεώσεων για τη συμμόρφωση με διατάξει διεθνού προστασία και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζητούμε περισσότερε κατευθυντήρε γραμμέ για τον εντοπισμό και την παραπομπή ε, ατόμων που χρήζουν διεθνού προστασία. Αυτό πρέπει να είναι μέσα στον επιχειρησιακό προγραμματισμό όλων των κοινών επιχειρήσεων ε, του ε, Frontex. Επίση, θα καλωσορίζαμε μία αναφορά στα πρότυπα που υπάρχουν μέσα κατευθυντήρε γραμμέ σχετικά με τι αρχέ τη μη επαναπροώθηση στα πλαίσια των συντονισμένων θαλασσίων θαλασσίων επιχειρήσεων του Frontex. Επίσης, προτείνουμε ο προβλεπόμενος κώδικας συμπεριφοράς και ο ανεξάρτητος μηχανισμό παρακολούθησης που προβλέπονται για τις διαδικασίες επιστροφή να αναπτυχθεί και να υλοποιηθεί και για το προσωπικό του Frontex και για τους συνοριοφύλακες που εμπλέκονται σε όλες τις κοινέ επιχειρήσεις και σε όλα τα πιλωτικά προγράμματα. Διάφορες τροπολογίες αποσκοπούν στην ενίσχυση των ικανοτήτων του Frontex, ούτως ώστε να αντιδρά καλύτερα στι στις προκλήσεις σχετικά με τον συντονισμό και τη διαχείριση ε, των δράσεων ε, για τα εξωτερικά σύνορα. Τονίζουμε όμω ότι η ενίσχυση του Frontex ε, που δεν είναι πρέπει να παρακολύσει, το αντίθετο πρέπει να διευκολύνει του παρατηρητέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αιτούν άσυλο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάρτιση είναι για κέρια σημασία, ε, κοινό υλικό για την κατάρτιση. Αυτό έχει απασχολήσει το Frontex τα τελευταία χρόνια. Καλωσορίζουμε τι προτάσει σχετικά με βάσει των οποίων θα πρέπει όλο το προσωπικό που εμπλέκεται σε επιχειρήσει ε, να καταρτίζεται σχετικά με την διεθνή προστασία και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, υπάρχει αναφορά σε ειδικέ οργανώσει, οργανώσει προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναφέρονται ως ενδυνάμει εταίροι του Frontex ε, για την ανάπτυξη περαιτέρω διδακτικών εργαλείων. Επίσης, ε, στις κοινέ ε, ομάδες ε, υποστήριξη καλούνται τα κράτη-μέλη να τηρούν τις βασικές υποχρεώσεις ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και αναφέρεται συγκεκριμένα η αίτηση ασύλου. Σε αυτά τα μέτρα, η πρόταση της Επιτροπής αφορά στις κοινέ επιχειρήσεις, στις συντονισμένες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερο συντονισμός, καλύτερη παρακολούθηση και καλύτερη αξιολόγηση. Καλωσορίζουμε αυτές τις νέες διατάξεις, αλλά θεωρούμε ότι η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων περί προστασία. θα πρέπει να είναι εκ των ονού κάνευ ε, ε, για τον τερματισμό μιας επιχείρησης ε, του Frontex. Επίση, συγκεκριμένη αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και στι υποχρεώσει περί διεθνού προστασία στι τακτικέ εκθέσει που θα υποβάλλονται από τον Frontex και προβλέπονται μονάδε εμπειρογνωμόνων. Η κυρία Λοχπίλερ το αναφέρει στη γνωμοδότησή τη. Μπορεί να έχουν κέριο ρόλο τέτοιε ομάδε εμπειρογνωμόνων. Τέλο, θα προτείναμε επίσης ε, περαιτέρω αναφορά σχετικά με το άσυλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή να ζητήσουμε ανεξάρτητη αξιολόγηση από ομάδε εμπειρογνωμόνων, ε, ε, είτε επί τούτο είτε δυνάμει φυσταμένων διατάξεων, και σε σχέση με το ρόλο της, ε, του Frontex ε, για τις διαδικασίες επιστροφής αναγνωρίζουμε το δικαίωμα των κρατών μελών να επιστρέφουν άτομα ε, τα οποία μετά από δίκη η εξέταση του αιτήματό τους κρίνεται ότι δεν χρειάζονται διεθνή προστασία αλλά τονίζουμε ότι αυτές οι επιστροφές θα είναι βιώσιμες μόνο αν γίνουν σε εθελοντική βάση και υλοποιούνται με τρόπο ώστε να υπάρχουν προοπτικές ουσιαστικής επανένταξης αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία προέλευσής τους. θέλουμε να έχει ενισχυμένο ρόλο Frontex στις κοινέ επιχειρήσεις της επιστροφής, ε, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν τα για και τα ελάχιστα πρότυπα ε, που προβλέπουν μεταξύ άλλων στην οδηγία της επιστροφής, ε, δηλαδή συγκατάθεση για την υποχρεωτική επιστροφή και περιορισμός της βίας που επιτρέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Συγγνώμη κυρία Γκάρλικ, μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα, με να μπορείτε να επιβραδύνετε και δεν έχουμε και πολύ χρόνο, αλλά μην μιλάτε φυσικά πιο γρήγορα τώρα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Όχι, όχι, όχι, θα, θα, θα κλείσω για να ακούσουν και άλλες φωνές. Τέλος, ε, πιστεύουμε ότι η αιτήσια έκθεση για τις διαδικασίες επιστροφής του Frontex και κυρίως ως προς τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να κοινοποιούνται, να δημοσιεύονται προς όφελος του Κοινοβουλίου και άλλων θεσμικών οργάνων που παρακολουθούν τις δραστηριότητες του Frontex. Συνεχίζουμε να έχουμε δέσμευση για συνεργασία με το Frontex και θα επικουρούμε παρέχοντας συμβουλές ε, το Frontex κάθε φορά που οι δραστηριότητες του Frontex έχουν ε, επίπτωση σε άτομα τους οποίους ε, καλούμε να προστατεύσουμε. Σας ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε τώρα εν συντομία τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, ο κύριος Νίλσεν. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σε ευχαριστώ για τη δυνατότητα που δίνετε να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση. Η δυνάμωση της πτυχής ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κανονισμό Frontex ήταν μία από τις κύριες προτεραιότητες της ε, Επιτρόπου μάλιστα όταν είπε αυτή την πρόταση και γι' αυτό χαίρομαι για την θετική υποδοχή της οποίας έτυχε αυτή μας η πρόταση. Σύντομα, με δύο λόγια να υπάρχει κάποια καλύτερη παρουσίαση του ρόλου του Frontex τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τον την κοινωτική νομοθεσία και το χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν ελέγχουν τα εξωτερικά τα εξωτερικά σύνορα. Έχουμε 900 εκατομμύρια, 900 εκατομμύρια διαβάσεις από τα ευρωπαϊκά σύνορα κάθε χρόνο. Όλος ο Frontex εδώ είναι και θα είναι πολύ περιορισμένος. Frontex δεν μπορεί να συμμετάσχει λειτουργικά στις διαδικασίες αυτές στα σύνορα. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να δούμε ότι πραγματικά ποσοτικά οι παρεμβάσει Frontex είναι πολύ περιορισμένε και θέλω να σα υπενθυμίσω ότι είτε είναι παρόν είτε όχι το Frontex. Το ίδιο πλαίσιο νομικό για την, με την κοινοτική νομοθεσία και τη χάρη των ανθρώπων δικαιωμάτων πρέπει να εφαρμόζεται. Θα μπορούσα να πω να εφαρμόζεται με τα υψηλότερα ε, ε, με τις πρώτες αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά δεν το λέω γιατί ή εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται. Δεν είναι θέμα ποσοτικής εφαρμογής. Στο ρόλο του Frontex θα πρέπει να αναλάβει τη δική του ευθύνη σαν δημοσιαρχή και να αναλάβει ε, τις ευθύνες για τη συμβολή στην πλήρη συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διάρκεια των ε, διαδικασιών που συντονίζει. Δεν μπορεί όμως να πάρει εκείνο την ευθύνη και να μειώσει την ευθύνη των κρατών μελών. Το κύριο θέμα που είναι δύσκολο, παραδέχομαι, είναι ποιος είναι ο αποδεκτός ρόλος του Frontex. όταν το λέμε αυτό είναι ότι δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ε, Frontex σαν μια υπηρεσία λήψης αποφάσεων. Η άρνηση ενδεχομένω ε, εισόδου σε εκείνους που ζητούν το άσυλο είναι πάντα αρμοδιότητα και ευθύνη των κρατών μελών. δεν μπορούμε ο ε, Frontex να είναι ο δημόσιος κατήγορος ή ο δικαστής. Αναφερόμενο σε ορισμένε από τι παρατηρήσει που έγινε είναι ότι πραγματικά θα πρέπει τα στοιχεία για τα γεγονότα που ε, έχουν παρατηρηθεί θα πρέπει να ισχύουν και για την ε, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι σαφέ αυτό. Frontex θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ε, βάλει τέρμα ε, στη διαδικασία αυτή σε περίπτωση που υπάρχει παρεμβίωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να έχουν πάντα τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες για όλους τους ε, εμπλεκόμενους και όλοι οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι δημόσιοι. Δύο λόγια για τα προσωπικά στοιχεία. Αυτή τη στιγμή ο Frontex προωθεί, επεξεργάζεται πραγματικά ανθρώπινα, ε, συγγνώμη, ε, προσωπικά στοιχεία για τους ανθρώπους που έχουν περάσει από το σύστημα αυτό. Η Κομισιόν δεν προτείνει κάτι διαφορετικό στη νέα εντολή για το Frontex, αλλά είναι κάτι που θα συζητήσουμε μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Άσυλο. τονίζω την ανάγκη να υπάρχει καθαρός διαχωρισμός μεταξύ του Frontex και της νέας υπηρεσίας ασύλου όσον αφορά τις αρμοδιότητες. Από την άλλη μεριά όμως είναι αναγκαία η στενή συνεργασία. Το είπαμε αυτό πάντα ξεκάθαρα. Ιδανικά θα θέλαμε τα κράτη-μέλη να υποστηρίζονται λειτουργικά από τη Frontex, από τις ε, συνολικές υπηρεσίες και από τη νέα υπηρεσία για το άσυλο. Τελευταία παρατήρηση, Πρόεδρε, με την άδειά σα, το θέμα τη ε, παρακολούθηση των κοινών ε, δραστηριοτήτων. Δεν θα είναι την στο γεγονό ότι η συμμετοχή παρατηρητών στι διαδικασίε αυτέ προβλέπεται από τι προτάσει και θα πρέπει να ε, έχουμε κατά νου την υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων για τους πρόσφυγες. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον πρόσωπο του Frontex, ο κύριος Μπάγκνερ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που δίνετε στο Frontex να λάβει το λόγο στη συζήτηση αυτή. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Νίλσεν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημεριζόμαστε την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Καταρχήν, να σας πω πόσο Frontex λαμβάνει υπόψη το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις δραστηριότητες του. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Λόχ Πίλερ ότι όπως και ε, ο ΙΕ και οι οργανισμοί του ΙΕ, ο Frontex θα πρέπει να τηρεί και να εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διαχείριση, του, στη διαχείριση των συνόρων. Αυτό είναι βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής διαχείρισης των συνόρων. Είναι προφανές άλλωστε ότι ο Frontex δεν είναι πολιτικό όργανο και οι δραστηριότητες του στον τομέα αυτό θα πρέπει να εντάσσεται στις ε, σχέσεις συνεργασίας που έχουμε με τις κοινωτικέ χώρες αλλά και με τρίτες χώρες. Οπότε αυτήν την άποψη θέλουμε η διάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων να διαπνέει όλες τις ε, δραστηριότητές μας, τις ε, κοινέ επιχειρησιακές δραστηριότητες ή το capacity building. Φυσικά δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την προσπάθεια. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε υποστήριξη των στρατηγικών μας εταίρων όπως είναι η Πατιαρμοστία και οι άλλοι οργανισμοί του ΟΗΕ αλλά ταυτόχρονα να εμπλέξουμε και τα κράτη-μέλη στη στρατηγική που θέλουμε να διαμορφώσουμε ώστε και, τα κράτη, ότι, ώστε και εμείς να συμπεραλάβουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις δραστηριότητες συνεργασίας που έχουμε. Αναφέρθηκε η έλλειψη λογοδοσίας, η έλλειψη διαφάνειας. Πρόθεση μας πάντως είναι να συστήσουμε και ένα διοικητικό συμβούλιο που θα είναι ανοιχτό και στο οποίο θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και θα είναι ανοιχτό και προς ε, τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και προς τις αρχές συνοριοφυλάκων, ώστε να καταρτήσουμε ένα κοινό σχέδιο παρακολούθησης για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια. Τώρα για να δούμε πώς ο σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει συμπεριληφθεί στις δραστηριότητες του Frontex, θα ήθελα να πω ότι στην ανάλυση κινδύνων που πραγματοποιούμε προσπαθούμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το άσυλο και το Σύμφωνο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η ανάλυση κινδύνων είναι σημείο φετηρίας των δραστηριοτήτων μας προκειμένου να προσαρμόσουμε τις αντιδράσεις μας και την επέμβασή μας στο θέμα σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εδώ είναι πολύτιμη συνεργασία που έχουμε με την υπατερμοστία γιατί από εκεί αντιλούμε πολλές πληροφορίες για ροές ετούντων ασύλου από τα εξωτερικά σύνορα και σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήρες γραμμές έχουμε συζητήσεις με την ΆΣΟ αλλά και με την υπατερμοστία Αρμοστία του ΟΗΕ, γιατί αυτό περιλαμβάνεται και στο σύστημα της Στοκχόλμης το πεδίο συνεργασίας μεταξύ Frontex και ASO για, την, για τον εντοπισμό ετούντων άσυλο. 1,5 λεπτό σας έχει απομείνει γιατί ήδη έχουμε υπερβεί το ωράριό μας. Καλώς, καλώς. Θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Frontex θα πρέπει με διεθνείς κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες που Φυσικά περιλαμβάνει και το θέμα του σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αυτό αναφέρθηκε και στι κοινέ μα δραστηριότητε. Το ανέφερε αυτό ο Έλληνα Ευρωβουλευτή. Χρειαζόμαστε συμφωνία και διαβούλευση και με το συμμετέχον κράτο, αλλά και με το κράτο πρόλευση. Δεν μπορούμε εμεί να επιβάλλουμε συγκεκριμένε δραστηριότητε στα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε συνεργασία μαζί του. Σε ό,τι αφορά την κατάρτιση, φυσικά θέλουμε να καλύψουμε όλη την κοινότητα συνοριοφυλάκων. Έχουμε κοινές, ε, ε, κοινά σεμινάρια, ειδικευμένους ε, εταίρους και σε ό,τι αφορά τη σχέση με τις τρίτες χώρες, αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της εντολής μας που θα διαβριθεί και περαιτέρω και είναι μια κατάσταση αρκετά περίπλοκη και δημιουργεί προκλήσεις γιατί φυσικά θα έχουμε συνεργασία και με τις εθνικές υπηρεσίες συνόρων των τρίτων χωρών, αλλά ταυτόχρονα με, τις, με τη συνεργασία που έχουμε θα προσπαθήσουμε να φέρουμε οριζόντια και πάντα παρούσα στην συνεργασία μας τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Και τώρα ο κύριος Ζέμκε, ο αντιπρόσωπος και μετά θα ξανακούσουμε την εισηγήτρια ο αντιπρόεδρος κύριο Ζέμκε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά, αλλά δυστυχώ έχουμε πρόβλημα γιατί μα έχει απομείνει ελάχιστο χρόνο και ο κανονισμό για το Frontex είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και όχι μόνο ο κανονισμό, και η γνωμοδότηση τη υποεπιτροπή μα έχει τεράστιο βάρο και ελπίζω θα γίνει δεκτή και θα ληφθεί υπόψη από την ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή τη γνωμοδότηση της κυρίας Λοχμπίλερ και έχουν υποβληθεί 21 τροπολογίες. Ε, όπως μας συνηθίζει η κυρία Λοχμπίλερ και πάλι κατάρτισε πολύ μεστή πρόταση και συμφωνώ με το 90% περίπου των τροπολογιών σας και των προτάσεών σας κυρία Λοχμπίλερ. Φυσικά δεν συμφωνώ 100% μαζί σας. Κατά την γνώμη μου υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η επέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με ποιο βαθμό θα μπορούσαμε να ελέγξουμε τις δραστηριότητες του Frontex. Κατά τη γνώμη μου, σε ορισμένες περιπτώσεις ε, είμαστε υπερβολικοί και το παρατραβάμε κατά τη γνώμη μου ότι αφορά αυτή την επέμβαση. Και θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην τροπολογία σας υπαριθμών 20... Έχετε βέβαια πολύ καλές προθέσεις και συμφωνώ με τις καλές σας προθέσεις, αλλά νομίζω ότι το παρατραβάτε κυρία Συγήτρια. Για παράδειγμα, εδώ πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να ασχοληθεί και με όλους τους με όλες τις διατάξεις τις ε, λεπτομεριακές και τις οργανωτικές στη σχέση με τις τρίτες χώρες. Γιατί έχουμε 27 χώρες και οι διατάξεις όταν έχουν απλώ οργανωτικό χαρακτήρα, σημαίνει ότι κάθε τρει και λίγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ασχολείται με πολύ λεπτομεριακέ και πολύ αποσπασματικέ διατάξει που αφορούν τι σχέσει του οργανισμού με τι χώρε αυτέ. Νομίζω ότι εδώ το παρατραβάμε ω προ το εύρο του ελέγχου. Επαναλαμβάνω κυρία Λόχμπιλερ, στο 90% των περιπτώσεων έχετε απόλυτο δίκιο, οι προθέσει σα είναι πολύ αγαθέ, αλλά μερικέ φορέ. Είστε λίγο υπερβολικοί και σχολαστικοί και χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της σχολαστικότητας και είναι η τροπολογία 20. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ακούσαμε επαρκή υποστήριξη για την έκθεση της εισηγήτριας και από την Κομισιόν και από τη Φρότεξ. Θα δούμε λοιπόν πώς θα προωθηθεί αυτή η γνωμοδότηση στις επόμενες εβδομάδες όταν θα υποβάλουν και οι συνάδελφοι τροπολογίες και θα περάσει την πρώτη Δεκεμβρίου στην ΑΦΕΤ. Ίσως μπορεί να παρουσιάσει τα γλίγορα τα τελευταία της σχόλια, εισηγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους και θα προσπαθήσω να λάβω υπόψη όλες τις παρατηρήσεις που έγιναν Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που με επένεσαν ότι εργαστικά πραγματικά εις βάθος. Αυτό δεν οφείλεται στην ε, ε, εθνικότητά μου, αλλά επειδή έχουμε τώρα μια κατάσταση όπου μπορούμε κάτι να καθορίσουμε, πράγμα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε προηγουμένως. Και χαίρομαι που τώρα η Frontex δεν λέει όχι, δεν θα εργαστούμε πάνω σε αυτό, αλλά ακούσαμε ότι υπάρχουν σκέψεις να υπάρχει μια ειδική και η ετήσια έκθεση και μια έκθεση παρακολούθηση. Γι' αυτό ήμουν ένα εις βάθος, γιατί πραγματικά η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σημαντική στις λεπτομέρειες και μπορούμε να δούμε πώς θα πρέπει να τροποποιήσουμε, αλλά στο Κοινοβούλιο υπάρχει μια ομάδα εργασία που ασχολείται γενικά με τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς μπορούν να ληφθούν υπόψη για τις περαιτέρω εργασίες του Κοινοβουλίου. Βέβαια, θα ήθελα να συνεχίσω να συνεργάζομαι και με τον κύριο Πορσίνη και με τον συνάδελφο από τη Λίμπε. Έχουμε τους ίδιους στόχους, αλλά αυτό το παράδειγμα ότι θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των σκέψεων για την ασφάλεια αφενός και τα ανθρώπινα δικαιώματα αφετέρου δεν είναι ένα επιχείρημα που μου αρέσει, γιατί αυτό σημαίνει ότι όταν έχουμε λιγότερη προσέγγιση των δοκιμάτων έχουμε περισσότερη ασφάλεια. Ίσως δεν το εννοείται έτσι, αλλά θα ήθελα να το πω ξεκάθαρα. Όταν έχουμε μία δράση όλων των διαφορεμένων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα έχουμε περισσότερη ασφάλεια τελικά, όχι λιγότερη. Και θα ήθελα να σα υπενθυμίσω, όχι μόνο με τη Frontex, αλλά γενικά ε, για τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζει τα σύνορα της Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν ε, σεβόμαστε ανθρώπινα δικαιώματα θα έχουμε προβλήματα αξιοπιστίας έναντι άλλων περιοχών. Κατά πόσο πραγματικά να πάμε σοβαρά υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και λοιπόν θα δώσω ένα παράδειγμα. Ε, θεωρούμε ότι από τότε που άρχισε να, να εργάζεται η Frontex, όχι μόνο η Frontex, περίπου 60.000 ε, άτομα ε, συνελήφθησαν στη θάλασσα γιατί ε, παραβίασαν σύνορα. Και αυτή την ερώτηση που τι έγινε με αυτά τα άτομα, η απάντηση ήταν «Ε, μα δεν είναι μόνο η Frontex που συμμετείχε εκεί στις συλλήψεις αυτές, αλλά ε, δεν ξέρουμε καθόλου τι έγινε με τα άτομα αυτά. Δεν ξέρουμε αν επαναπατρίστηκαν ή τι. Ζητώ συγγνώμη, θα συνεχίσουμε στα αγγλικά αν το επιτρέπετε. Ε, είναι έκτακτες συνθήκες. Εντάξει, θα προσπαθήσω. Η υπόλοιπη συνεδρία θα διεξαχθεί δυστυχώς ε, στα αγγλικά.